Ε, Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Έχουμε την παρουσίαση της μελέτης της ΤΟΑ με θέμα τη γλωσσική ισότητα στην ε, ψηφιακή εποχή και το σχέδιο για μια ανθρώπινη γλώσσα. Ε, εξαιρετική έκθεση και μεγαλεπίβολο αυτό το σχέδιο προς μια ανθρώπινη γλώσσα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό παρουσία των μελών της Επιτροπής Πολιτισμού. Κάμερεβερτ. Η κυρία Κάμερεβερτ, που είναι η νέα πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, I hope to continue the good... με την οποία ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε την αγαστή μας συνεργασία. Ζητά συγγνώμη για την απουσία της. Οπότε θα ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης της ΣΤΟΑ που ενδιαφέρει τα μέλη και των δύο επιτροπών και της Επιτροπής Ήτρα και της Επιτροπής ΚΑΛΤ. Θα γίνει μια διεξοδική επισκόπηση της κατάστασης των τεχνολογιών ανθρώπινης γλώσσας, HLT. Πρόκειται για συστήματα λογισμικού που στόχο έχουν ε, να, καλύψουν την ανθρώπινη γλώσσα σε όλες τις μορφές, ε, γραπτή, προφορική και νοηματική. Και να δούμε ποιες είναι οι μελλοντικέ προκλήσεις ε, στον ευρωπαϊκό κλάδο της τεχνολογίας της ανθρώπινης γλώσσας. Το HLT και ίσως ε, μας βοηθήσει και έχει σημασία η τεχνολογία αυτή και για το μέλλον στην μετάφραση και στην διερμηνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, θα πρέπει να δούμε τον οικονομικό αντίκτυπο που έχουν οι γλωσσικοί φραγμοί στην Ευρώπη και ποιε είναι οι κοινωνικέ συνέπειε αυτή τη έλλειψη ισότητα που υπάρχει ε, τη τεχνολογική στήριξη όλων των ευρωπαϊκών ε, γλωσσών. Αλλά φυσικά ο δρόμο μπροστά μα είναι μακρύ Ίσως μετά από 15 χρόνια φτάσουμε σε τέτοιες γενικευμένες τεχνολογίες, αλλά σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει 24 επίσημες γλώσσες και πάνω από 60 γλώσσες μειονοτήτων και περιφερειακές, θα πρέπει να μπορούμε να επικοινωνούμε ε, διασυνοριακά σε όλες τις γλώσσες. Ε, αυτό, αυτή την πολυτέλεια θα πρέπει να έχουν οι πολίτες που μετακινούνται. Γιατί σκεφτείτε ότι στην Κίνα 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα, μπορούν να μετακινούνται ε, σε απέραντες εκτάσεις, ε, καταλαβαίνοντας ε, σχεδόν πλήρως τους συμπολίτες, τους Κινέζους, γιατί μιλούν την ίδια γλώσσα. Έτσι θα, με μια τέτοια προσπάθεια και ξεπερνώντας τους γλωσσικούς φραγμούς, θα φέρουμε πιο κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες, θα προωθήσουμε και την οικονομία μας και θα αξιοποιούμε καλύτερα τις ε, ευκαιρίες της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Έχετε λάβει τη μελέτη της ΣΤΟΑ και θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Ο εκπρόσωπος της ΣΤΟΑ, ο κύριος Ριβέρα, ε, έγκριτος εμπειρογνώμων και συντάκτη τη σχετική έκθεση. Ένα δεκάλεπτο, παρακαλώ, έχετε. Ευχαριστώ, κύριε Μπούζεκ, για την εισαγωγή και σα ευχαριστώ όλου που ήρθατε για να συζητήσουμε σήμερα αυτό το κρίσιμο για την Ευρώπη θέμα. Η, το τμήμα της ΣΤΟΑ εκπώνησε αυτή τη μελέτη με θέμα τη συνέπειες των γλωσσικών φραγμών στην Ευρώπη υπό το πρίσμα των τεχνολογιών ε, τη ανθρώπινη γλώσσα, προκειμένου να αξιοποιήσουμε την πολυγλωσία στην Ευρώπη στην ψηφιακή εποχή. Θα εξετάσουμε μια γκάμα θεμάτων σήμερα. Καταρχήν, την πολυγλωσία στην Ευρώπη και το πώ ε, οι φραγμοί γλωσσικοί επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία τη Ευρώπη. Δεύτερον, το, η θέση για το καθεστώ των τεχνολογιών ανθρωπιστική γλώσσα, οι μελλοντικέ τάσει αυτών των τεχνολογιών. Το τρίτο θέμα θα είναι κλάδος ε, των τεχνολογιών ανθρώπινης γλώσσας ε, στη βιομηχανία και στη, στη, στον κλάδο της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και οι διάφορες ε, ευκαιρίες και επιλογές πολιτικής που έχουμε στο τομέα των τεχνολογικών αυτών. Η Ευρώπη με 28 επίσημες γλώσσες και πάνω από 60 εθνικές, περιφερειακές και γλώσσες ε, έχει την πολυγλωσσία ως βασικό της πλούτο, βασικό στοιχείο της πολιτισμικής πολυμορφίας. Βλέπετε το χάρτη με τις γλώσσες και τη διαλέκτου στην Ευρώπη. Αυτή η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί όμως και από έναν από τους πιο σημαντικούς γλωσσικούς φραγμούς για τη δημιουργία μιας πραγματικά ολοκληρωμένης Ευρώπης στην ψηφιακή ε, εποχή. Πάνω από το 60% των Ευρωπαίων, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν την αγγλική, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν στα αγγλικά και υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και εντός των χωρών. Σε μερικές χώρες πάνω από 80% του πληθυσμού δεν δύναται να επικοινωνήσει στα αγγλικά στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ενώ το 20% του πληθυσμού δεν γνωρίζει τα αγγλικά στην Ολλανδία. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα σενάριο με τις έξι πλέον ομιλούμενε γλώσσες στην Ευρώπη, αυτές είναι τα ισπανικά, ε, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, πολωνικά και ισπανικά και 15% των Ευρωπαίων μένουν πίσω και 11%, των Ευρω... 11 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το μισό πληθυσμό δεν μπορούν να μιλήσουν σε αυτές τις πλέον ομιλούμενε γλώσσες. Βλέπετε τι μεγάλη διαφορά υπάρχει. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο γλωσσικό χάσμα που έχει ε, κοινωνικά και ε, δημογραφικά χαρακτηριστικά. Εξαρτάται ε, από το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών αν μιλούν αγγλικά ή όχι. Μάλιστα, όσο περνάμε την, ε, την ηλικία των 19 ετών ε, και έχουμε πανεπιστημιακές σπουδές, ε, κοσοπλασιάζεται η πιθανότητα να ξέρει κανείς ξένες γλώσσες. Οπότε υπάρχουν ε, πολλοί παράγοντες, γεωγραφικός, δημογραφικός και μορφωτικός. Και έχουμε σημαντικό τέτοιο γλωσσικό χάσμα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Ε, κοινωνική ένταξη των μεταναστών, ε, κινητικότητα των εργαζομένων, διεθνέ εμπόριο, διασυναριακό εμπόριο. Για παράδειγμα, με, στο θέμα το, της κινητικότητας των εργαζομένων, το ποσοστό των πολιτών που έχουν ε, μεταβεί σε άλλη χώρα για να διαμείνουν ή να εργαστούν είναι μόνο 6%. Η γλωσσική φραγμή είναι ο βασικότερος λόγος αυτού του χαμηλού ποσοστού των μετακινούμενων πολιτών. Και μάλιστα η ανάλυση δείχνει ότι θα αυξηθεί, αν δεν είχαμε του γλωσσικού φραγμού, θα είχαμε τριπλάσιο αριθμό συμπολιτών μα που θα μετέβαιναν σε άλλη χώρα για να παραμείνουν ή να εργαστούν, αν δεν υπήρχαν οι γλωσσικοί φραγμοί. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Υπάρχει μεγάλο κατακαιρματισμό τη αγορά αυτή τη στιγμή, ε, στις, ε, ανάλογα με τι πολιτισμικές και γεωγραφικέ. Ε, ε, ιδιότητες. Επίσης, ε, στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή ο αριθμός των πολιτών που κάνουν ε, online αγορές είναι μηδενικός. Αν δεν είχαμε τέτοια γλωσσικούς φραγμούς, οι Ευρωπαίοι πολίτες που θα ψώνιζαν ηλεκτρονικά στην Ουγγαρία θα αυξανόταν και θα φτάνουν μέχρι τα 6 εκατομμύρια, που είναι τριπλάσιος αριθμός από αυτό που τώρα ε, αγοράζουν ηλεκτρονικά από την Ουγγαρία, που είναι σήμερα 2,2 εκατομμύρια. Για τις χώρες αυτές ήταν τεράστια επιτυχία η υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών, γιατί θα γίνονταν πιο ανταγωνιστικές τέτοιες χώρες που είναι σήμερα απομονωμένες και θα είχαν περισσότερο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το θέμα είναι πώς οι τεχνολογίες ε, της γλώσσας μπορούν να συμβάλλουν στην ε, υπέρβαση αυτού του γλωσσικού φραγμού. Καταρχήν έχουμε πολλές ψηφιακές ε, εφαρμογές, ψηφιακή συνδρομή όπως ε, το High Cortana και επίσης έχουμε διάφορα τμήματα, το έξυπνο περιεχόμενο, διαδραστική, διαδραστικός λόγος και μηχανική ή αυτοματοποιημένη μετάφραση, που είναι σημαντικότερος ε, τρόπος για να υπερβούμε το γλωσσικό φραγμό. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη και πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα και γι' αυτό οι τεχνολογίες ε, της ανθρώπινης γλώσσας θα μπορέσουν να αποτελέσουν πραγματική λύση για την υπέρβαση του ε, γλωσσικού φραγμού. Δεν χρειάζεται να καταλάβετε αυτό το, την περίπλοκη εικόνα, αλλά η Google λέει ότι πλησιάζει πια να φτάσει την ανθρώπινη ποιότητα κατά την πραγματοποίηση μεταφράσεων, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Οπότε στο εγγύς μέλλον θα αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες και θα μπορέσουν πια να προσφέρουν πραγματικά ποιοτικέ φάμιλε τη ανθρώπινη μετάφραση από υπολογιστέ. Τέτοιου είδου τεχνολογίε βέβαια στηρίζονται στα δεδομένα, οπότε χρειαζόμαστε αρκετά δεδομένα μεταξύ των διαφόρων γλωσσών για να λειτουργήσουν αυτέ οι τεχνολογίε. Γιατί αυτέ οι τεχνολογίε βασίζονται στη χρήση τεράστιων ε, ε, ε, ποσοτήτων δεδομένων. Και μάλιστα στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη διαφορά της γλωσσικής υποστήριξης ε, ε, των τεχνολογιών. Είχαμε μία μελέτη πριν από μερικά χρόνια που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι για τις περισσότερες γλώσσες το επίπεδο στήριξης για τις περισσότερες ήταν είτε πολύ χαμηλό είτε ανύπαρκτο. Και αυτό οδηγεί όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως ε, λιγότερο ομιλούμενες, σε έναν ψηφιακό αφανισμό που θα ήταν σημαντικό πρόβλημα για την Ευρώπη. Τώρα, ο κλάδος ε, των τεχνολογιών αυτών ε, ανθρώπινης ε, γλώσσας είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το οικοσύστημα, το ίντερνετ, κυριαρχείται κυρίως από μη ευρωπαϊκές εταιρείες, μεγαθύρια. Και εκεί τα αγγλικά είναι η βασική γλώσσα στο οικοσύστημα του ίντερνετ. Βλέπετε την πράσινη γραμμή που είναι η στήριξη στην αγγλική γλώσσα και η στήριξη που έχουν άλλες γλώσσες στο οικοσύστημα του διαδικτύου. Ε, περίπου 500 εταιρείε ε, στην Ευρώπη έχουμε που σχετίζονται με τις τεχνολογίες αυτές. Ένα τέταρτο είναι πολύ μικρές, μόνο 6% είναι μεγάλες τέτοιες εταιρείε. Οι περισσότερες πάντως είναι επιχειρήσεις με λιγότερο από 200 ε, εργαζομένους και ένα τέταρτο επαναλαμβάνουν πολύ μικρές επιχειρήσεις με πολύ λιγούς στο πολύ δεκά εργαζόμενους. Και μια και ψάχνουμε το οικοσύστημα, η Ευρώπη έχει μια μακρά παράδοση έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με πάνω από 800 τέτοια κέντρα. Και μάλιστα είχαμε πολύ επιτυχημένα σχέδια στην Ευρώπη, όπως το MOSES, που το χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βιομηχανία που είναι ένα λογισμικό μετάφρασης μηχανικής ε, ανοιχτού κώδικα και διευκολύνει τη μετάφραση σε πολλές γλώσσες. Βέβαια το οικοσύστημα τη έρευνα στην Ευρώπη δυστυχώ έχει αποτύχει στην προσπάθεια να κινητοποιήσει επενδύσεις σε τέτοιου είδου τεχνολογίες. Οπότε είναι τεράστιες οι προκλήσεις για τον ε, κλάδο αυτό. Μεγάλος κατακαιρματισμός. Οι βασικοί παράγοντες ε, είναι κυρίως αμερικανικές εταιρείες. Ακόμη και οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, έχουν εξαγοραστεί από μεγάλες ε, αμερικανικές πολυεθνικές που κυριαρχούν σε αυτό το τοπίο του διαδικτύου. Η Ευρώπη ε, έχει κάποιε ερευνητικέ δραστηριότητε, αλλά είναι μεμονωμένε. Οπότε χρειαζόμαστε πολύ ισχυρότερο συντονισμό των δικών μα πρωτοβουλειών, των ευρωπαϊκών. Θα πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, ε, να αυξήσουμε την ε, τεχνογνωσία και την κοινή διαχείριση και να αναβαθμίσουμε τι ευρωπαϊκέ εταιρείε και να επενδύσουμε και στι υποδομέ και στου πόρου μόνο με την αναβάθμιση αυτών των επιχειρήσεων μπορούμε να έχουμε και στην Ευρώπη ισχυρέ πολυεθνικέ ευρωπαϊκή ε, ιδιοκτησία. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με τι πολιτικέ μα είδαμε ότι οι τεχνολογίε ανθρώπινη γλώσσα είναι πολύ σημαντικέ για την Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον και τέτοιου είδου τεχνολογίε θα μα επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει. Οπότε θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Έχουμε αναλύσει πάνω από 3.000 ε, τεχνικά, πολιτικά, στρατηγικά εγγραφά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορε αναρτήσει και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερω απογοητευτικά. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα ε, στη σύγκριση του πώς ε, ε, καλύπτουν αυτά τα έγγραφα θέματα όπως είναι υπολογιστική, το διαδίκτυο των αντικειμένων ή τεχνολογίες της ανθρώπινης γλώσσας. Πολλά από τα έγγραφα αυτά οι μπλοκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου δείχνουν ότι ένα πολύ μικρό τμήμα τους αφιερώνεται σε αυτές τις τεχνολογίες. Είναι σχεδόν ανύπακτες. Το ίδιο φαίνεται και από τα έγγραφα πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, στην, στην στρατηγική της ενιαίας ψηφιακής αγοράς του 2015 υπάρχει μία σύντομη μόνο παραπομπή στις πολυγλωσσικές υπηρεσίες. Ενώ είδαμε στην μελέτη μας ότι η γλωσσική φραγμή είναι από τους σημαντικότερους φραγμούς της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Μας εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι παρά το ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα των τεχνολογιών, δεν ε, τη της προσοχής από τα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Τώρα, προτείνουμε κάποιες θεσμικές πολιτικές για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, να γίνει μια σωστή αξιολόγηση των πολιτικών και να προταθούν ερευνητικές πολιτικές για την ενίσχυση και τη στοχευμένη έρευνα από τι τεχνολογίε ανθρώπινη γλώσσα για να προωθήσουμε τη δημιουργία ευρωπαϊκών πλατφορμών, όχι μόνο για τα αγγλικά, αλλά και για τι μικρότερε ε, γλώσσε τι λιγότερο ομιλούμενε, ώστε να γεφυρώσουμε αυτό το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσών. Επίση, ε, προτείνουμε και πολιτικέ για την αγορά για να συνειδητοποιηθούν οι πολίτε, οι εταιρείε, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί για το πώ μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί επειδή δεν αντιλαμβάνονται πολύ ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χορηγήσουν ε, πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον όπως η Ευρώπη. Θέλουμε επίσης να υπάρξουν ε, δημόσιες ή μικτές επενδύσεις και θερμοκοιτίδες για να βοηθήσουμε αυτές τις εταιρείες. Επίσης, πρέπει να υπάρξει περισσότερη κατάρτιση προσωπικού για τα θέματα αυτά. Και προτείνουμε και μερικές ε, δημόσιες πολιτικές, για παράδειγμα, να υπάρξουν τέτοιες δημόσιες υπηρεσίες ε, στην Ευρώπη σε πολλές γλώσσες και να στηρίξουμε και τον κλάδο στην Ευρώπη. Ε, με συγχωρείτε που μιλάω πολύ γρήγορα. Αυτά είναι τα θέματα και ποια είναι τα πορίσματα. Η γλωσσικοί φραγμή είναι πολύ σημαντική στην Ευρώπη και έχουν πολύ ισχυρέ και οικονομικέ επιπτώσει. Οι τεχνολογίε ε, τη ανθρώπινη γλώσσα ε, αναπτύσσονται πολύ γρήγορα με βάση αυτά τα ε, δίκτυα νευρώνων. Έχουμε δυνατότητε να υπερβούμε αυτού του φραγμού με τι νέε τεχνολογίε. Ο κλάδο δεν μοιάζει να κάνει πολλά για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός και από πλευράς ε, πολιτικών δεν ε, αντανακλώνται αυτά τα θέματα στην πολιτική πληροφορική της Ένωσης. Αυτό είναι αναπάντεχο και προτείνουμε να υπάρξουν πολιτικές ε, επιλογές πολιτικής για να διορθώσουν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος για την παρουσίασή σας. Να καλωσορίσω θερμότατα τον συνάδελφο που είναι πρώην μέλος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας, τον Βιτόριο Πρόντι. Σε ευχαριστώ Βιτόριο για την παρουσία σου. Σε θυμόμαστε πολύ καλά, τουλάχιστον οι παλαιοί. Και είστε πάντα ιδιαίτερα καλοδεχούμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Ήσασταν ιδιαίτερα ενεργό μέλος της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, want to say Αν θέλετε να πείτε κάτι, ε, με χαρά να σας ακούσουμε. Κύριε Πρόεδρε, με συγκινείτε. Επανέρχομαι μετά από δυόμιση χρόνια σε αυτό το θεσμό που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και στην κατανόηση που απέκτησα των προβλημάτων της ανθρωπότητας και της ε, οικονομίας. Εξακολουθώ να εμπνέομαι από αυτό το πνεύμα του οποίου έγινα κοινωνός κατά τη σχέση μου μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους και πρώην συναδέλφους εδώ, σε αυτό το χώρο που ήταν τόσο σημαντική εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ Βιτόριο, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε θερμά. Δεν είμαστε πρώην συνάδελφοι, εξακολουθούμε να είμαστε συνάδελφοι. Είστε επισκέπτης μας, αλλά είστε πρώην μέλος. Λοιπόν, να περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος ε, Παουλ Ρίμπιχ. Ξέρετε, Βιτόριο, τίποτα δεν αλλάζει στην Επιτροπή μας. Ο Πάουλ είναι ε, πρόεδρος ε, της ομάδας μελέτης ΤΟΑ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που μου κάνατε. Η ΣΤΟΑ είναι ένας οργανισμός επιλογής των τεχνολογικών και επιστημονικών επιλογών. Βλέπουμε δηλαδή τι δυνατότητες θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον για να σημειώσουμε επιτυχίες ε, στην πολιτική μας, στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Και φυσικά το να καταλάβουμε οι μεν τους δε είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για να κάνουμε τη δουλειά μας και γι' αυτό μεταξύ των πέντε προτεραιοτήτων της ΤΟΑ πρώτον η διεθνή κινητικότητα ούτως ώστε να είναι βιώσιμη δεύτερον ε, η βέλτιστη χρήση των πόρων των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Τρίτον, να δούμε πώς αντανακλάται ο πραγματικός κόσμος ε, στον ιονή κόσμο, τον κόσμο της τεχνολογίας. Δεύτερον, πώς μπορούμε να θέτουμε στην ε, διάθεση των ανθρώπων της τεχνολογίας, για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας. Ας πούμε ότι είστε σε ένα αεροπλάνο και έχετε ένα πρόβλημα υγείας και η γλώσσα σας δεν είναι πολύ διαδεδομένη. Πώς θα έχετε υπηρεσίες στη διάθεσή σα, ώστε σύντομα και αποτελεσματικά να μπορείτε να εξηγήσετε τι έχετε και τα μαζικά δεδομένα μας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις γλωσσικές δεξιότητες. Και αυτός είναι ένας ε, επιχειρηματικός κλάδος ε, με κύκλο εργασιών ε, στο μέλλον πολλών δισεκατομμυρίων. Είναι λοιπόν βασικό να ξεκινήσει κανείς από το νηπιαγωγείο. Και είχαμε πάει πέρυσι με το ΣΤΟΑ στην, στο Silicon Valley και το Google μας είπε ότι 1% των κερδών της εταιρείας αυτής δίδεται για κοινωνικούς σκοπούς, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, ε, για παράδειγμα ε, διένυμαν 500.000 iPhone, πήγαν εκεί στα hotspot με τους ε, πρόσφυγες και χρειάστηκε να επινοήσουν μια νέα βρόσα γιατί χρειάστηκε να δουν πώς θα μπορέσουν να συνεννοηθούν με ανθρώπους που δεν γνώριζαν παρά μόνο αραβικά. Ξεκίνησαν λοιπόν όπως οι Κινέζοι με ιδεογράμματα για να αναπτύξουν μια νέα βάση για μια νέα γλώσσα, για να μπορούν να συνοηθούν. Βλέπετε ότι στο ίντερνετ σήμερα πουλούνται όλα. Και όταν συζητάμε για το γεωμπλοκάρισμα στο ίντερνετ, βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχει ένας φραγμός από τη μία χώρα στην άλλη που είναι ο γλωσσικός φραγμός. Και για να μπορεί κανεί να είναι σε επαφή με την οικονομία, τον πολιτισμό και τέτοια, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει τη γλώσσα για να έχει μια ποιοτική επικοινωνία. Γι' αυτό προτείνω για το ένα το πρόγραμμα έρευνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που τώρα αρχίζουμε να εκπονούμε, να ε, συζητήσουμε και την γλωσσική ενιαία αγορά, να δημιουργήσουμε δηλαδή τι αναγκαίε υποδομέ, ούτω ώστε να υπάρξουν ε, ερευνητικέ εργασίε και επιστημονικές εργασίες για να διατηρήσουμε τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης. Έτσι νομίζω ότι θα αποκτήσουμε και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εδώ έχουμε για παράδειγμα 20 γλώσσες, τις οποίες ε, μελετάει κατόπιν ε, το Google και προσπαθεί να δει πώς είναι δυνατόν να φτιάξουμε φράσεις όλες αυτές τις γλώσσες. Νομίζω ότι η μετάφραση η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας κλάδος που πρέπει να ενισχύσουμε με τους αλγορίθμους που χρειαζόμαστε για να καταλαβαίνουμε και να γινόμεθα αντιληπτοί στον κόσμο. Αυτός ο, ο κόσμος λοιπόν της ε, τεχνολογίας μπορεί να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ο Σνάλφος Σαουντάργας, ο οποίος αυτός είχε κάνει την πρόταση για αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για αυτή την ε, πάρα πολύ καλή μελέτη, την οποία εκπώνησαν έμπειροι επιστήμονες και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη ΣΤΟΑ για την υποστήριξη αυτής της ιδέας. Δεν ε, θα σχολιάσω τη μελέτη αυτή καθεαυτή, διότι πρέπει να τη μελετήσουμε. Υπάρχουν πολύ καλές ιδέες, αλλά ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, τι έχει η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μια πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική κληρονομιά και μια καλή ε, πολιτική η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στις συνθήκες. Έχει εξαιρετικές δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό το οποίο δεν διαθέτει η Ευρώπη είναι μια πολιτική πολυγλωσσίας ε, και πολυπολιτισμικότητας ε, στον, στην εποχή της ε, ε, πληροφορικής. Δεν έχει πολιτική στον ψηφιακό χώρο για τις γλώσσες. Και σε αυτό υστερεί η Ευρώπη, όπως ε, ήδη αναφέρθηκε. Οι βασικές εξελίξεις στην τεχνολογία της γλώσσας γίνονται εκτός Ευρώπης. Η Ευρώπη κάνει πολλά, αλλά δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν διακαώς αυτή τη μελέτη και στη μελέτη αναφέρονται ήδη και κάποιες κατευθύνσεις των πολιτικών. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με στόχο μια ευρωπαϊκή πολιτική πολυγλωσία στην ψηφιακή εποχή. Και τέλος, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω ως παράδειγμα Αναφέρθηκε και το Google, είδαμε και στην οθόνη ε, πρόσφατα ότι υπήρξε πρόοδος ε, στο λεγόμενο δίκτυο βαθιάς ε, μάθησης και αυτά έγιναν στην Ευρώπη. Ε, η Google ε, απόκτησε την DeepMind, η οποία έδρευε στο Λονδίνο. Και υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα, προγράμματα της ανθρώπινης ε, τράπεζας, της Human Bank. Γιατί γίνονται λοιπόν όλα αυτά εκτός Ευρώπης και δεν γίνονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει απαντήσεις. Εγώ δεν είμαι κατά του προγράμματος αυτού, είμαι αναφανδόν υπέρ, αλλά πρέπει ε, ε, δεν θα έλεγα να, ε, να σπαταλήσουμε χρήματα, αλλά πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα και να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες κάπου συγκεκριμένα. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Υπάρχει το πρόγραμμα αυτό για την ανθρώπινη γλώσσα. Θα πρέπει να το προχωρήσουμε λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε το Human Language Project. Ίσως θα μπορούσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσουμε και κάποιο ψήφισμα για να το προεθήσουμε αυτό ευχαριστώ. κύριε Στουσιαντόφσκι. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια των προελισσάντων γιατί συμφωνώ μαζί τους. Πιστεύω και εγώ ακράδαντα ότι η βασική πρόκληση αυτής της μελέτης είναι να δούμε πώς θα ερμηνευτεί ε, και πώς θα αξιοποιηθούν αυτές οι νέες τεχνολογίες και τα μαθηματικά μοντέλα και οι αλγόριθμοι. Mm. Γιατί δεδομένη της ε, γλωσσικής μας πολυμορφίας και της πολιτισμικής μας πολυμορφίας που αποτελούν τμήματα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, mm. μας ενδιαφέρει να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό είναι για μας, για την Ευρώπη, από ε, για την Αμερική που δεν έχει τέτοιους γλωσσικούς φραγμούς ούτε τόσο μεγάλη γλωσσική πολυμορφία. Εμείς όμως με τη γλωσσική πολυμορφία μας ε, δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η πιο σημαντική γλώσσα. Όλες οι γλώσσες είναι ισότιμες και ο πλούτος μας έγκυται σε αυτή την πολιτισμική πολυμορφία και σε γλώσσες που μιλούνται εδώ και αιώνες. Έχουμε εδώ μια μαθηματική ερμηνεία αυτού του κλάδου των τεχνολογιών της ανθρώπινης γλώσσας και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε διάφορες μεθόδους για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και να ξεπεράσουμε τους γλωσσικούς φραγμούς. Και συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να παραμελούμε αυτό το κλάδο. Να μην θεωρούμε ότι η κατάσταση ε, είναι δεδομένη, ότι ε, πολλοί είναι γλωσσομαθείς και ότι δεν χρειαζόμαστε τέτοιες τεχνολογίες. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε πολύ πιο εντυπωσιακέ ε, τεχνολογίες και η πρόοδος είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από ό,τι στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να ανασκουμποθούμε και να δούμε τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε εμείς αυτά τα θέματα. Έχουμε λύσεις ε, στα πλαίσια της μηχανικής αυτοματοποιημένης μετάφρασης ε, Θα πρέπει να δούμε πώς μελετάμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο και από εκεί και πέρα να δούμε τι τεχνολογίες μας εξυπηρετούν περισσότερο. Πάντως θα πρέπει να ξεχνούμε και τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τον τρόπο λειτουργίας του, γιατί αυτή η μελέτη θα μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο σε πολλούς το... τομείς ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ, κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη θαυμάσια παρουσίαση και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Παύλο Ρούμπιχ και τη ΣΤΟΑ που ε, παρήγγειλαν αυτή τη μελέτη και ε, τον Σνάλφο Σαουντάργας που την πρότεινε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο Σαουντάργας ο οποίο εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με το θέμα της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη και πάντα τονίζει ότι το θέμα αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο των ε, εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πρώτη παρατήρηση. Η γλώσσα για μένα είναι τμήμα του πολιτισμού. Χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει πολιτισμός. Η Ευρώπη ζει από την ε, πολιτιστική της πολυμορφία. Οπότε αυτά τα οποία μας είπατε εδώ είναι πολύ βασικά. Πρέπει οπωσδήποτε η γλωσσική μας πολυμορφία να διατηρηθεί στην Ευρώπη. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Άρα δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε. Δηλαδή να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό, να διατηρήσουμε σε υψηλή θέση παντού όπου έχουμε δυνατότητα ο καθένα τη γλώσσα του και κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε, κάτι που υπερβαίνει το πλαίσιο τη έκθεσή σα. Το θέμα είναι πώ μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, ούτω ώστε αυτή η γλωσσική πολυμορφία να προωθηθεί, να ευνοηθεί πολύ περισσότερο, όπω ακριβώ είπε και ο συνάδελφο. Αυτό νομίζω πρέπει να επιχειρήσουμε. Δηλαδή δεν αρκεί να λέμε ότι α, τι άσχημο που είναι που παίζει τόσο ισχυρό ρόλο η αγγλική γλώσσα στο ίντερνετ. Να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Ούτω ώστε να διατηρήσουμε τη γλωσσική και πολιτιστική μας πολυμορφία. Δηλαδή και μέσω των νέων μέσων και μέσω των νέων τεχνολογικών εξελίξεων να αξιοποιηθούν περισσότερο όλες αυτές οι γλώσσες. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ίσως κάποια άλλη μελέτη μέσω της ΤΟΑ. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε. Ούτως ώστε να ευνοήσουμε ακόμη περισσότερο την ε, γλωσσική πολυμορφία. Στις 23 του Ιουνίου βέβαια πέρυσι η Βρετανία αποφάσισε να αποχωρήσει. Όταν θα προκύψει λοιπόν το Brexit θα πρέπει να δούμε το γλωσσικό μας καθεστώς, πώς θα το διαμορφώσουμε, αν θα πρέπει να το τροποποιήσουμε και σε τι βαθμό θα έπρεπε να αποδώσουμε μεγαλύτερο ρόλο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε άλλες γλώσσες. Αλλά εντάξει, α δούμε τώρα πώ θα προχωρήσει το Brexit και μετά το δούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιάρομιρ Κόχλιτσεκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή υπάρχει διερμηνία, θα μιλήσω κι εγώ στη μητρική μου γλώσσα, την τσεχική δεν ε, ξέρω σε ποιο βαθμό ιστό εξετάζει και διάφορες οικογένειες γλωσσών και το γεγονός ότι κάποιες οικογένειες γλωσσών χρησιμοποιούν αντίστοιχη σύνταξη. Σε όλες τις ε, μεταφραστικές μηχανές υπάρχει πάντα η δυνατότητα ε, μετάφρασης άρθρων από εφημερίδες ή άλλων γραπτών κειμένων, αλλά μόλις ε, υπάρχει κάποιο κείμενο ιδιαίτερα τεχνικό, ε, διαπιστώνει κανείς κάποιες συγκεκριμένες εκφράσεις ε, για τη συγκεκριμένη επιστήμη μπορεί, ή τέχνη. Μπορεί να είναι η αλλουργία, μια επεξεργασία μεθόδων ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται λοιπόν για ε, αντικείμενα τα οποία είναι δύσκολα. εγώ ε, ε, είμαι από αυτούς που ε, κάνουν επιμέλεια μεταφράσεων για να ελέγξουμε κατά πόσον η τεχνική ορολογία που χρησιμοποιείται είναι σωστή. Και πρέπει να φροντίσουμε ταυτόχρονα να είναι σωστή η σύνταξη, η διατύπωση, αλλά επίσης να είναι και σωστό το κείμενο από τεχνικής σκοπιάς. Και αυτό φυσικά ε, είναι κάτι που ακόμα δεν μπορούν να κάνουν μεταφραστικέ ε, μηχανές. Ευχαριστώ. Ναι και, ναι και μιλούμε για πολυγλωσία σήμερα. Θα πρέπει τουλάχιστον σήμερα να μιλάμε όλη τη μητρική μας γλώσσα. Εγώ θα προσπαθήσω να συνεχίσω να μιλάω πολωνικά. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον κύριο Μάρκο Μαρτσέλα, από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Θα σας παρακαλούσα όμως να είστε εξαιρετικά λακωνικός, Στο πολύ ένα λεπτό, όχι παραπάνω, γιατί μας περιμένουν έξω οι Μαλτέζοι Υπουργοί. Χαίρομαι πάντως που δίνει το παρόν στη συνεδρία σε αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρακαλώ ένα λεπτό το πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη ΣΤΟΑ για την έκθεση αυτή και ε, αναγνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες ε, για να ε, προωθήσουμε το ρόλο της τεχνολογίας για να άρουμε τους γλωσσικούς φραγμούς και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτών των διαφορών λόγω γλωσσικών φραγμών. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε ότι ακόμα και από τεχνικούς ε, ε, τρόπους είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες πηγές γλωσσών. Είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που δίνονται ε, μέσω τεχνολογίας και έρευνες, ε, κυρίως για τα μηχανήματα αυτόματης μετάφρασης και τα συστήματα μάθησης, τα νευρονικά δίκτυα ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και θα τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς θα μπορούσατε να μιλήσετε τη μητρική σας γλώσσα. Αλλά εντάξει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα γνωρίζετε βέβαια. Ο κύριος Λάγκεν, ο επόμενος ομιλητής. Ε, Είμαι υπέρ της μελέτης αυτής. Είμαι εδώ και 23 χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω διαπιστώσει πως Ακόμη και εμείς οι ίδιοι δεν εκφραζόμεθα στην γλώσσα μας και την υποτιμούμε. Βλέπουμε πόσο κυριαρχεί στις συζητήσεις ε, η αγγλική γλώσσα και πολλές φορές μας δημιουργεί δυσχέρειες με διάφορες τεχνικές έννοιες. Και εμείς ε, που είμαστε αρμόδιοι συνομοθέτες πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε έναντι της διοίκησης να τους τονίζουμε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι γλώσσες. Αν πάει κανείς στη Washington σε ένα μουσείο, στο Μουσείο Διαστήματος για παράδειγμα, κάθε έκθεμα αναφέρεται σε τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες, δηλαδή περιγράφεται αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά και αγγλικά. Ενώ εδώ μέσα μόνο αγγλικά μιλάμε και καμιά φορά και λίγα γαλλικά. Οι άλλες ε, σημαντικές γλώσσες, ε, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πολωνικά, εξαφανισμένες. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η έκθεση γιατί και εμεί πρέπει να ξαναδούμε τι κάνουμε εδώ πέρα μέσα. Ιδιαίτερα όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει, θα μα μείνουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν τα αγγλικά ως επίσημη γλώσσα, αλλά η μεγαλύτερη από πλευρά εκπροσώπηση σίγουρα δεν θα είναι πλέον η αγγλική γλώσσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λάγκεν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μερικές φορές ξεχνάμε τις μητρικές μας γλώσσες, αλλά κάπως θα πρέπει να συνεννοούμαστε και στους διαδρόμους όταν συναντιόμαστε. Δεν έχουμε συνέχεια δίπλα μας διερμηνείς, οπότε δεν έχουμε άλλη λύση με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρούμε μια κοινή ε, ε, γλώσσα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εδώ βέβαια στη συνεδρίαση τα πράγματα είναι προφανή και έχει δίκιο, μπορούμε να μιλάμε όλη τη γλώσσα μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εμπειρογνώμονά μα ε, για μια σύντομη, σύντομη παρακαλώ απάντηση, γιατί ελάχιστο χρόνο έχει μείνει. Μα περιμένουν, όπω σα είπα, έξω από την αίθουσα υπουργοί. Well, thank you very much. Um, I think... Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σήμερα ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για τις γλώσσες μας και πώς θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε όταν συνομιλούμε και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό νόημα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε πολλές γλώσσες και ο καθένας θα πρέπει να μιλάει τη μητρική του γλώσσα και να μπορούν να ε, μιλούν τη γλώσσα τους ε, όταν ε, αποτείνονται και σε δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη. Αυτό έπρεπε να είναι το πολιτικό θεματολόγιο της Ευρώπης, αλλά μέχρι τώρα δεν, έχει καταφέρει, δεν έχουν καταφέρει να βρουν μια λύση, γι' αυτό η Αγγλική έγινε η γλώσσα εργασίας της Ευρώπης. Τώρα όμως είναι η ευκαιρία. Με την εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών έχουμε αυτή την τεχνολογία. Και νομίζω ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να κάνει αυτά τα κρίσιμα κρίσιμα βήματα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε θερμά και περιμένουμε και τη συνέχεια της ε, έκθεσης, μια επόμενη μελέτη προς την ίδια κατεύθυνση φυσικά. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο υπαριθμών 12,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 Uh, and gentlemen. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, περνάμε στη συνάντησή μας με την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάλτα. Θα μιλήσουμε για τις προτεραιότητες της πολιτικής τηλεπικοινωνιών και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο κύριος ε, Εμμανουέλ Μαλέια είναι ο Μαλτέζος Πρωθυπουργός για τον, ε, υπουργός, συγγνώμη, για, τον, την ανταγωνιστικότητα ε, και τις ψηφιακές και ναυτιλιακές υπηρεσίες. Και έχουμε και τον κύριο Κρίς Ατζούς. Ατζούς, Ατζούς. Ο αρμόδιος κοινοβουλευτικός γραμματέας για την έρευνα, την καινοτομία, την νεολαία και τον αθλητισμό. Θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας στα θέματα έρευνας, καινοτομία και διαστήματος. Πολύ σημαντική για μας αυτή η συζήτηση. Θα θέλαμε να μιλήσουμε και για τον ΕΝΙΣΑ, την ενιαία ψηφιακή αγορά, τη, την οικονομία των ψηφιακών αυτιλιακών υπηρεσιών, την ανταγωνιστικότητα, το GRC, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, η IT, η ITER. Αν θέλετε μπορείτε να μας μιλήσετε και για αυτά τα θέματα, γιατί έχουν αναγγελθεί ως προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ένα άλλο θέμα είναι η πρωτοβουλία Πρίμα, που συζητήσαμε το πρωί. Έχουμε επίσης το νέο κώδικα τηλεπικοινωνιών και την υπόθεση της ε, περιαγωγής στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής. Πολύ σημαντικά θέματα. Θα ακούσουμε την παρουσίασή σας και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω θερμότατα τους υπουργούς από τη Μάλτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή μας είναι, είναι αρμόδια για όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα, την πολιτική τηλεπικοινωνιών, την ενία ψηφιακή αγορά. Οπότε, ίσως θα μπορούσα να ζητούσα πρώτα από τον ε, Υπουργό Μαλέια να μας κάνει την παρουσίαση και μετά θα περάσουμε στον συνάδελφό του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ καταρχάς στο γενικότερο πρόγραμμα της Προεδρίας της χώρας μου, στα Μαλτέζικα, και στη συνέχεια θα περάσω στην αγγλική γλώσσα για τις προτεραιότητές μας. Στη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών η Ευρώπη, 60 ε, ετών, η Ευρώπη ήταν το σύμβολο της ειρήνης, της ανάπτυξης και της ελπίδας. Και αυτό φυσικά ήταν λόγω των πρωτοπόρων του ευρωπαϊκού οράματος, όταν ε, πολλοί άλλοι ήταν επιφυλακτικοί και είχαν δισταγμούς όσον αφορά το πόσο επιτυχημένοι μπορούμε να είμαστε και αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Στην 60 επέτειο του Ευρωπαϊκού Οράματος επαφείται πλέον σε εμά, τη Μάλτα, το μικρότερο κράτος μέλος, να έχουμε την ευκαιρία και την ε, δυνατότητα να προεδρεύουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια ε, χρονική στιγμή που θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα τελευταία 60 χρόνια. Έχουμε όλοι καθήκον να προστατεύσουμε όσα έχουμε αποκτήσει μέχρι τούδε και να ε, μεταλαμπαδεύσουμε τα ωφέλη αυτά στους πολίτες μας. Οφέλη, τα οποία ορισμένες φορές λησμονούμε αποτελεί επίσης και χρυσή ευκαιρία προκειμένου να ατενίσουμε το μέλλον. Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα όθηση και οι πρόσφατες εξελίξεις ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πολύ πιο κοντά στους πολίτες της και ε, να ε, διαβιβάζει τα μηνύματά της με πιο αποτελεσματικό τρόπο για τα μέτρα στήριξης τα οποία λαμβάνει προκειμένου να παράσχει καλύτερες ευκαιρίες στους πολίτες της για να τους δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους και να είναι επιτυχημένοι. Οι πολιτικές εξελίξεις που βιώσαμε την περασμένη χρονιά ε, μας έχουν σημαδέψει όλους. Η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις ε, δεν ήταν ποτέ τόσο επίγουσα και η έκκληση να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες μας ποτέ δεν ήταν πιο σαφής. Οι εξελίξεις ε, την τελευταία χρονιά έφεραν τριγμούς στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μάλτα είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο ευρωπαϊκό όραμα. Ελπίζουμε ότι στη διάρκεια της Προεδρίας μας, χάρη στη δουλειά μας στο Συμβούλιο και στη συνεργασία μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, αποβίνει κίτρια και να είναι ισχυρότερη. Ξέρουμε ότι έξι μήνες είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ε, και παρά το γεγονός ότι φιλοδοξούμε ε, και θέλουμε να προωθήσουμε αρκετά προγράμματα και να είναι και πιο αξιόπιστα, είμαστε και ρεαλιστές. Γνωρίζουμε τι περιορισμούς έχουμε και γνωρίζουμε επίσης και τι μπορούμε να κάνουμε και ποια είναι τα ισχυρά μας σημεία. Ε, θα προσπαθήσουμε λοιπόν ε, να προχωρήσουμε με τους συνομιλητές μας στο Συμβούλιο χωρίς ε, να κρύψουμε τίποτα και χωρίς κρίνες προθέσεις. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πνεύμα συνεργασίας και ειλικρίνειας. Το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό μα και ο αναπληρωτή Πρωθυπουργό, ο Υπουργό Οικονομικών και ο επικεφαλή τη αντιπολίτευση έχουν όλοι διατελέσει μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σημασία που έχει. Ε, εσείς είστε οι άμεση εκπλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να νομοθετείτε προ το συμφέρον του. Είναι τιμή μα να προεδρεύουμε στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τέτοια χρονική στιγμή. Ο φάρος που θα μας καθοδηγήσει ε, στα διάρκεια της Προεδρίας μας είναι να δώσουμε μια νέα όθηση σε οτιδήποτε βοηθήσει τους πολίτες να έρθουν πιο κοντά σε εμά ως καταναλωτές, ως άνθρωποι που δημιουργούν πλούτο και ως ενδιαφερόμενοι. Επομένως, γι' αυτό το λόγο ε, έχουμε καθορίσει τις έξι προτεραιότητες. Μετανάστευση, ασφάλεια, ε, πολιτική γειτονία, κοινωνική ένταξη και ε, ναυτιλιακά ζητήματα ως ε, τις βασικές μας προτεραιότητες, διότι θεωρούμε ότι οι χώρες μας ε, έχουν πολύ σημαντικές ανησυχίες για τα θέματα αυτά. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ ε, ενδελεχώς σε κάθε προτεραιότητα, αλλά με την άδειά σας κύριε Μπούζεκ ε, θα αναφερθώ στο πρόγραμμα εργασίας, στους τομείς που συζητά η δική σας η Επιτροπή και που αφορούν και τις δικές μου τις αρμοδιότητες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους για τη θερμή υποδοχή είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι προσκεκλημένος στην Επιτροπή Ήτρε για να παρουσιάσω τις ψηφιακές προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Από τότε που ανέλαβα καθήκοντα ως Υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων έχω αναλάβει να προσπαθήσω να συναντηθώ με όσο το δυνατόν περισσότερους από εσά. Οι συναντήσεις αυτές επέτρεψαν και σε μένα και στην ομάδα μου να αντιληφθεί ποιες είναι οι προτεραιότητες και ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ψηφιακά ζητήματα. Ανέκαθεν πίστευα ότι το να υπάρχει ένας ανοιχτός και ειλικρινός δίλαυλος επικοινωνίας με τον συνομιλητή μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι γνώμονας επιτυχίας της Προεδρίας μας. Και σας διαβεβαιώ ότι εμείς από την πλευρά μας σκοπεύουμε να κρατήσουμε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς στη διάρκεια όλης της Προεδρίας μας ως ε, νησιωτικό κράτος ε, που δεν έχει χερσαία σύνορα με την υπόλοιπη Ευρώπη, ε, αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά τα ωφέλη της διασύνδεσης και της ψηφιοποίησης. η αυγή της ψηφιακής εποχής ε, μας οδήγησε σε μια εποχή γεμάτη νέες ευκαιρίες, οι οποίες, ε, ε, δεν θα μπορούσαμε, τις οποίες δεν θα μπορούσαμε καν να τις διανοηθούμε πριν από κάποια χρόνια και θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε όχι μόνο να ολοκληρώσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά, αλλά επίσης να δώσουμε και μάχη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε θα επιτύχουμε αρκεί όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για τα επόμενα επόμενα χρόνια. Γι' αυτόν τον λόγο και σε στενή συνεργασία και με τους εταίρους μας από την Τρόικα, το Τρίο των Προεδριών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Μάλτα θέλει να ξεκινήσει και να προσπαθήσει να υλοποιήσει ένα ρεαλιστικό θεματολόγιο στη διάρκεια της Προεδρίας της. Η Μαλτέζικη Προεδρία θα συνεχίσει το πολύτιμο έργο που έκαναν η Ολλανδική και η Σλοβακική Προεδρία, τα μέλη του Τρίου των Προεδριών, και να διασφαλίσει ότι το επόμενο τρίο θα έχει και ισχυρά θεμέλια επί των οποίων θα οικοδομήσει τι πολιτικές του. Όσον αφορά την, ε, την τεχνολογία 5G, επειδή είναι ε, πρώτων πυλών, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται ε, στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και το Connecting Europe μπορεί να δώσει εξαιρετικές ευκαιρίες για το μέλλον. Η Μαλτέζικη Προεδρία θα προσπαθήσει λοιπόν να συνεργαστεί και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις ε, για τις ε, συχνότητες 470-490 ε, MHz ε, αποτελούν παράδειγμα της πολύ καλής συνεργασίας που θέλουμε με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έργο για τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα αποτελέσει και ε, μεγάλο τμήμα των εργασιών της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ε, το έργο για τον κώδικα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Μαλτέζικη Προεδρία θεωρεί ότι ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για, τις, τον τομέα των τηλεπικοινωνιών που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και τις μελλοντικές προκλήσεις και εξελίξεις εντός του ψηφιακού κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Μάλτα θεωρεί ότι εάν μπορέσουμε να έχουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα βασίζεται σε αυξημένη διασύνδεση και καλύτερους κανόνες ε, θα ε, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Γι' αυτό και ακριβώς συνεχίσαμε το έργο για τον κώδικα και προσπαθούμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε στενή συνεργασία και με τη μελλοντική Εστονική Προεδρία, αλλά και με τον εισηγητή αρμόδιο για το θέμα αυτό, για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα όσο περισσότερο μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να επανεξετάσουμε την πρόοδο ε, στο ε, Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών στις 9 Ιουνίου του 2017. Η Μαλτέζικη Προεδρία θέλει επίσης να ολοκληρώσει και την όλη αναθεώρηση του θέματος της περιαγωγής. Ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς και είμαι πεπισμένος ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρους, προκειμένου να έχουμε ένα νέο καθεστώς περιαγωγής μέχρι τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος. Οι διαπραγματεύσεις και από τις δύο πλευρές ε, είναι δύσκολες από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά είμαι πεπισμένος ότι και οι δύο πλευρές έχουν το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας επί του ζητήματος. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς περιαγωγή θα αποτελέσει ε, βοήθεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ε, βλέπουμε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Η Μαλτέζικη Προεδρία επίση σκοπεύει να ολοκληρώσει τον κανονισμό για την προώθηση τη σύνδεση στο διαδίκτυο στι τοπικέ κοινότητε και σε δημόσιου χώρου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξ όσων γνωρίζουμε, θα έχει ολοκληρώσει την εσωτερική του διαδικασία τον Απρίλιο. Και θα ήθελα να σα ε, καθησυχάσω και να σα πω ότι θα είμαστε και εμεί έτοιμοι να ξεκινήσουμε τριμερείς διαπραγματεύσει επί του ζητήματο με σκοπό να το ολοκληρώσουμε. Η Μαλτέζικη Προεδρία επίσης ε, θα ε, ε, συμπέσει και με την ε, επέτειο των δύο ετών της έναρξης της ψηφιακής στρατηγικής. Ε, θα κάνουμε έναν απολογισμό των ε, νομοθετικών ε, ζητημάτων που έχουμε και θα δούμε και τη στρατηγική μας. Η Μάλτα σκοπεύει η Προεδρία αυτή να είναι μια επιτυχημένη Προεδρία για όλη την Ευρώπη. Εάν συλλογικά καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε πλέρως την νέα ψηφιακή αγορά, θα έχουμε απτά ωφέλη για τις οικονομίες μας τις επιχειρήσεις μας και τις οικογένειές μας θα άρουμε φραγμούς για το εμπόριο και θα βελτιώσουμε την προστασία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Αξιότιμα μέλη, ως Προεδρία η πρόθεσή μας είναι να εργαστούμε αποτελεσματικά και αποδοτικά προκειμένου να επιτύχουμε τον κοινό στόχο της διαμόρφωσης της Ευρώπης σε ένα ε, ηγετικό ρόλο και θα βρίσκεται τα ψηφιακά θέματα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, ε, της ασφάλειας ε, προς το συμφέρον των πολιτών μας και των επιχειρήσεών μας. Δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε μόνοι μας αυτό. Για να μπορέσουμε πραγματικά να επιτύχουμε τους στόχους μας, ε, θα χρειαστούμε και τη στήριξη και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε ευγνώμονες για αυτή τη συνεργασία και Είμαστε βέβαιοι ότι από κοινού μπορούμε να προσφέρουμε μια καλύτερη Ευρώπη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Minister. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Και τώρα, έρευνα, καινοτομία και διάστημα. Ο κύριος Κρίς Άτζους, που είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά, για την έρευνα την καινοτομία, την νεότητα και τον αθλητισμό. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σα, ε, αξιότιμα μέλη. Σα ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου που είμαι εδώ ενώπιον σα για να σα παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασιών τη ε, Προεδρία τη Μάλτα στον τομέα τη έρευνα, τη καινοτομία και του διαστήματο. Η Προεδρία μα κατανοεί τη σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είναι οι συνομοθέτες. Και δεσμευόμεθα για ένα ανοιχτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε λοιπόν να χαιρετήσουμε τη σημασία αυτής της ανταλλαγής απόψεων. Όπως ξέρετε η Μάλτα ανέλαβε την εναλλασσόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά μετά την ένταξή της την 1η Μαΐου του 2004. Η Προεδρία της Μάλτας ε, θα λάβει η χώρα σε μια πολιτική συγκυρία ιδιαίτερα σημαντική για την ε, πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωσή μας. Θεωρώ ότι στον τομέα της έρευνας ανάπτυξη του διαστήματος θα συμβάλλουμε ουσιοδός ούτω ώστε να προωθήσουμε μια σειρά από θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την ε, σχέση μας με τις βασικές προτεραιότητες ε, των περιοχών γειτονία Ευρώπης και ιδιαίτερα την προώθηση του ναυτιλιακού τομέα για την έρευνα και την καινοτομία. Θα ασχοληθούμε με δύο θέματα. Να προχωρήσουμε τη συζήτηση για το πρίμα, την εταιρική σχέση για την έρευνα και καινοτομία στην ε, περιοχή της Μεσογείου, από τη μία, και την ορθο, τον εξορθολογισμό της υποβολής εκθέσεων. Πρώτα απ' όλα το πρίμα θα ασχοληθεί με τα τρόφιμα και τη διαχείριση των υδάτων για να επιχειρήσει να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια επενδύσεων στον, στην περιοχή της Μεσογείου. Θα αξιοποιήσουμε ως βάση το άρθρο 185 για να προωθήσουμε εταιρική σχέση για πρώτη φορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, χωρών της Μεσογείου που δεν ανήκουν στην Ένωση. Για πρώτη φορά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο κατέτοιο να συνεχιστεί η ανάπτυξη και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, γειτονία της. Το πρίμα είναι έκφραση του θεματολογίου του Επιτρόπου Μουέντας για να είμαστε ανοιχτοί προς τον κόσμο και για να έχουμε έμπρακτη επιστημονική διπλωματία. Η επιστήμη και η διπλωματία θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην πρόθεση των διεθνών σχέσεων και ιδιαίτερα για να αντιμετωπίσουμε μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις που από την ίδια τους τη φύση είναι φυσικά διαμεθοριακές. Η έναρξη αυτή, αυτού του σχεδίου για πρώτη φορά με το άρθρο 185 σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι για ορισμένα θέματα θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε κοινό έδαφο. Αλλά στόχο μα είναι να προχωρήσουμε με τη βοήθειά σα για την νομοθετική πτυχή του θέματο, ούτω ώστε να καταλήξουμε στην ε, εφαρμογή του προγράμματο πρίμα. Θα συνεργαστούμε λοιπόν στενά με την Επιτροπή Ήτρε για να προωθήσουμε το θέμα αυτό μέσω των αναγκαίων συζητήσεων και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει καλή θέληση από όλε τι πλευρέ σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο των διαφόρων κρατών για να επιτύχουμε του στόχου μα μέχρι το τέλο τη ε, Προεδρία μα. Τώρα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου προ την εισηγήτρια του πρίμα, την κυρία Σακοράφα, γιατί ανέλαβε την ευθύνη για να διατυπώσει την ε, άποψη της Επιτροπής σα, την έκθεση για το πρίμα. Από ό,τι καταλάβαμε, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεση έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στα πλαίσια των προσπαθειών της Προεδρίας να προωθήσουμε το θεματολόγιο για την ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας για την έρευνα και καινοτομία θα κάνουμε μια συνάντηση στη Μάλτα στις 4 ε, Μαΐου για να ενισχυθεί η συνεργασία στην ε, περιοχή μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και για να αξιοποιήσουμε την έρευνα ως μέσο για να καταλάβουμε τα βασικά αίτια της μετανάστευσης. Το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι η έγκριση μιας διακήρυξης της Βαλέτα για να ενισχυθεί η συνεργασία για την έρευνα και καινοτομία στον τομέα της Μεσογείου. Η δεύτερη προτεραιότητά μας αφορά την ε, επίβλεψη και την υποβολή εκθέσεων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Να δούμε δηλαδή που υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία μέσω πολλών εκθέσεων ούτω ώστε να εξορθολογήσουμε την προσπάθεια αυτή. Θέλουμε να απλοποιήσουμε την υποβολή εκθέσεων για τους ε, ασχολούμενους με την πολιτική έρευνα στην Ένωση. Θέλουμε οι ασχολούμενοι να βασίζονται σε στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων. Γι' αυτό η υποβολή εκθέσεων είναι απαραίτητη. Ωστόσο, χρειάζεται να κάνουμε υπερβολικέ εκθέσει. Γιατί αυτό δημιουργεί υπερβολική γραφειοκρατία. Και στην ουσία ε, δεν καθιστά δυνατή την εφαρμογή της πολιτικής μας. Θεωρούμε ότι οι υποχρεώσει υποβολή εκθέσεων με σωστό τρόπο θα επέτρεπαν ένα καλύτερο πλαίσιο πολιτική για περισσότερη αποδοτικότητα τη πολιτική μα στην έρευνα και καινοτομία. Στόχο μα λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για να δούμε διάφορε πλευρέ όπω η ισότητα και η συχνότητα των εκθέσεων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά οι Υπουργοί Έρευνας θα μπορούσαν να εγκρίνουν πορίσματα για να εξορθολογήσουν τη διαδικασία αυτή στο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνα στι 30 Μαΐου. Η Προεδρία μας επίσης δεσμεύεται να προωθήσει την εργασία που ξεκίνησε από το τρίο των ε, Προεδριών, δηλαδή να συνεχίσουμε τις συζητήσει για μια σειρά από επίκαιρα και πολύ σκόπιμα θέματα που αφορούν την πολιτική έρευνα τη Ένωση. Ένα τομέα που οπωσδήποτε θα είναι στο κέντρο της προσοχής μας είναι να κλείσουμε το χάσμα της καινοτομία. Δηλαδή μετά από την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την ειδική διάσκεψη για το θέμα αυτό κατά την ε, Σλοβακική Προεδρία. Το, η γεωγραφική ισορροπία για παράδειγμα στη συμμετοχή στο Horizon 2020 και στο επόμενο πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι προτεραιότητά μας. Διότι οπωσδήποτε ξέρουμε ότι και για σας είναι προτεραιότητα και σε σχέση με αυτό η Μαλτέζικη Προεδρία θα δει την δημοσίευση της πρώτης μελέτης επίπτωσης του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η Προεδρία μας γνωρίζει την ε, πολύ ουσιώδη δουλειά που έχει αναλάβει η Επιτροπή σας για να προπαρασκευάσει την επικείμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας. Χαιρετίζουμε αυτή την εργασία και προσβλέπουμε ε, στην δημοσίευση της έκθεσης της κυρίας Καπεθών Ρουίθ για την εφαρμογή του προγράμματος Horizon 2020 εν ώψη της ενδιάμεσης ε, αποτίμησης και των μελλοντικών προτάσεων για το ένατο πρόγραμμα. Η Προεδρία μας λοιπόν, στο μέτρο του δυνατού και σεβόμενη πλήρως ε, τις ε, ημερομηνίες, το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής, θα εργαστούμε για αυτή την ενδιάμεση αποτίμηση του προηγούμενου προγράμματος και θεωρούμε ότι φέτος θα καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις. Συνεργαζόμεθα λοιπόν με την επόμενη Προεδρία, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τη βάση για μια επιτυχημένη κατάληξη του θέματος αυτού. Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει δημιουργηθεί για να έχουμε συζητήσεις για διάφορα θέματα, θέματα καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Και θα σας καλωσορίσουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, της διοργάνωσης. Για παράδειγμα, η συστάση για την ανάπτυξη του, της μελλοντική ε, εμβληματικής πρωτοβουλίας για τις κβαντικές τεχνολογίες θα αποκαλυφθούν στη Μάλτα σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου για να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις για την επέκταση του προγράμματος για την ε, Μπλε Μεσόγειο σε μια ειδική εκδήλωση που θα γίνει στη Μάλτα στις 18 και 19 Απριλίου για θέματα τεχνολογίας. Θεωρούμε ότι η θαλάσσια έρευνα μπορεί να βοηθήσει για να έχουμε ένα καλύτερο ναυτιλιακό τομέα στην Ευρώπη. Επίσης θα έχουμε δύο άλλες ε, βασικές εκδηλώσεις για τις ε, ενέργειες Curie και άλλη μια εκδήλωση που θα γίνουν στις 11 και 12 Μαΐου και μεταξύ της 21ης και 23ης Ιουνίου αντίστοιχα. Τώρα, στον τομέα του διαστήματος θα εστιάσουν κυρίως οι συζητήσεις μας ε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής για μια στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα. Δημοσιεύθηκε τον περασμένο Οκτώβριο μετά από μια ευρεία και πλήρη διαβούλευση. Επειδή, όπως ξέρετε, αλλάζει το παγκόσμιο περιβάλλον, αναγνωρεί, γίνεται όλο και πιο ευρέω αναγνωρισμένη η στρατηγική σημασία του διαστήματος για την Ευρώπη. Άρα πρέπει να δράσουμε συλλογικά και ανεξάρτητα για να ε, είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας. Οι δραστηριότητες για το διάστημα βεβαίως είναι ζωτικές για την ανάπτυξη των κοινωνιών μας και έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό είναι ουσιώδες οι δράσεις μας να συνεχιστούν για να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες και το πλαίσιο για τις διαστημικές πολιτικές μας, να καθορίσουμε σαφείς στόχους στον τομέα αυτό για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να συμβάλλουμε σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη δυναμικού στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Κανένα μεμονωμένο κράτο μέλο ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, μεγάλο ή μικρό, μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο μεμονωμένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ενιαία στρατηγική για το διάστημα για να μεγιστοποιήσουμε τα θετικά ωφέλη από αυτή την πολιτική. Χαιρετίζω το γεγονό ότι η στρατηγική αυτή λαμβάνει υπόψη τι θέσει όλων των κρατών μελών καθώ και του Κοινοβουλίου μέσω των ψηφισμάτων, μέσω των ψηφισμάτων του για την ε, ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε από κοινού την προσπάθεια αυτή προ όφελο των πολιτών αλλά και του κλάδου στα πλαίσια αυτά. Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την ε, αντίδραση του Συμβουλίου σε αυτή την πρόταση. Και θέλουμε αυτό να γίνει Στι 30 Μαου στο Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα και το Διάστημα. Κατά την σε αυτή του Συμβουλίου θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για την εφαρμογή αυτή τη πολιτική διαδικασία αυτή θα προχωρήσει παράλληλα με την εργασία που κάνει η Επιτροπή σα για να διατυπώσει και την ε, στάση του Κοινοβουλίου. Και θα προκολουθήσουμε πολύ στενά αυτά που λέτε. επίση, είμαστε διατεθειμένοι να ε, αντιμετωπίσουμε και άλλε πρωτοβουλίε κατά την Προεδρία μα, συμπεριλαμβανομένε και τη προσπάθεια να ε, προωθήσουμε περισσότερο την ε, αγορά τέτοιων ε, δυνατοτήτων, δηλαδή να υπάρχει περισσότερη ε, συμμετοχή της οικονομίας στον τομέα αυτό. Και μαζί με τον Ευρωπαϊκό Φορέα για το Διάστημα θα οργανώσουμε μια διάσκεψη που θα έχει στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή της Μεσογείου σε αυτή την προσπάθεια στις 27 και 28 Ιουνίου. Θέλουμε να δούμε πώς οι τεχνολογίες του διαστήματος μπορούν να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από προκλήσεις, προκλήσεις στην περιοχή τη Μεσογείου που είναι μεγάλη σημασία για τη συνεχιζόμενη ασφάλεια και σταθερότητα της Ευρώπης. Το διάστημα θα συμπεριληφθεί επίσης και σε άλλες ε, τομεακέ εκδηλώσει. όπως για παράδειγμα η συνάντηση για την Μπλε Μεσόγειο που ανέφερα προηγουμένως. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένο ότι θα σας εμπνεύσει και στη δική σας εργασία το πρόγραμμα της Προεδρίας μας. Προσβλέπουμε στην επίτευξη με τη βοήθειά σας και τη συνεργασία σας αποτελεσμάτων, ούτως ώστε η Προεδρία μας να έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα προς το συμφέρον των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ. Ήδη ε, είχα πάει στη, για, Μάλτα για διακοπές. Τώρα αυτή τη φορά θα την ταυτίζουμε τη Μάλτα με, όχι ως ε, προορισμό διακοπών, αλλά ως ε, ε, χώρο διοργάνωσης πολλών εκδηλώσεων και συνεδριάσεων και άρα σκληρής εργασίας. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση εκ μέρους του ΕΛΚ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Καστίγια, Καστίγια Δεβέρα. Ευχαριστώ τη Μαλτέζικη Προεδρία και ευχαριστώ τους δύο υπουργούς που μας παρουσίασαν τις προτεραιότητες της Προεδρίας τους. Εγώ θα αποτωθώ κυρίως στον Υπουργό Μαλέγια, που είναι αρμόδιος για την πολιτική τηλεπικοινωνιών και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Είχαμε συναντηθεί και προηγουμένως, γιατί είμαι εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κώδικα για τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες και ξέρω πόσο πρόθυμος και συνεργάσιμος είναι ο υπουργό και ποιο είναι το ενδιαφέρον, το ζωηρό ενδιαφέρον της Μαλτέζικης Προεδρίας ε, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος και να διεκπαιρεωθούν ε, οι εκκρεμότητες σε αυτό το τομέα, οι ανοιχτές, τα ανοιχτά θέματα που μας έμειναν. Γιατί όλοι έχουμε επίγνωση της σημασίας που έχει η συμφωνία προκειμένου να ρυθμιστεί το, η περιαγωγή στην αγορά χοντρικής και στα μέσα Ιουνίου του 2017 είναι η διορία που έχουμε βάλει και τότε θα πρέπει να ε, καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής. Θέλουμε να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και είμαι βεβαίω ότι θα καταλήξουμε στη συμφωνία προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Πέραν του κώδικα των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών που με ενδιαφέρει και θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα. Έχουμε και άλλε νομοθετικέ πρωτοβουλίε σε αυτή τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών. Μία αφορά τον κανονισμό για το ασύρματο δίκτυο, το Wi-Fi, και είπατε ότι θέλετε στην Προεδρία σα ε, να καταλήξουμε σε συμφωνία και να μην ξεχνάμε και το BEREC, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, που επίσης ε, καλύπτεται από τη συνολική μεταρρύθμιση. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι επιτακτική ανάγκη της πρόοδου στο μέτρο του δυνατού. Μακάρι να μπορέσουμε στη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας να καταλήξουμε σε πολιτική τουλάχιστον συμφωνία για αυτή την πρόταση αναθεώρησης ε, της αγοράς ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε, αλλά αν μη τι άλλο να σημειώσουμε κάποια πρόοδο, γιατί και στο Κοινοβούλιο έχουμε επίγνωση της ανάγκης ε, πρόοδου στον κλάδο αυτό και μάλιστα με ταχύ ρυθμό. Γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον ψηφιακό κλάδο. Έχουμε ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, ελπίζουμε να το τηρήσουμε και αν όλα πάνε καλά θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά σύντομα, προς το καλοκαίρι. Πάντως, πιστεύω ακράδαντα ότι και το Συμβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν τη βούληση, την επιθυμία αλλά και την αποφασιστικότητα για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όποτε, οριμάσει, όποτε οριμάσουν οι συνθήκες, ώστε να έχουμε μια ποιοτική συμφωνία και φυσικά να μην καθυστερήσουμε και πολύ, γιατί είναι σχετικά επίγον το θέμα, όπως είπα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό Μαλέια και τον κοινοβουλευτικό γραμματέα Άτσους. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία προς τον Υπουργό Μαλέια για τον κώδικα τηλεπικοινωνιών που ανέφερε και η προλαλήσασα. Και να πω ότι τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κώδικα στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας στην εξέταση, αλλά και την αποτελεσματικότητα των παρόχων των υπηρεσιών, αλλά και των ε, ε, παρόχων υπηρεσιών δικτύου. Η, μια από τις πιο σημαντικές προτάσεις αφορά την εναρμόνιση των τιμών φάσματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμως βλέπουμε τις τιμές αυτές και σε ποιον χορηγήθηκε το φάσμα, βλέπουμε διαφορές, διακοιμάνσεις στις τιμές είναι πολύ διαφορετικές οι τιμές από χώρα σε χώρα. Όταν ε, βλέπουμε αυτές τις διαφορές, διαρωτόμαστε τι προτίθεται να κάνει η Μαλτέζικη Προεδρία για την νέα αυτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι στάση θα κρατήσει. Και προς τον κοινοβουλευτικό γραμματέα, τον κύριο Ατζούς, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προτεραιότητα του διαστήματος, αλλά να μην ξεχνούμε το γεγονός ότι η Μάλτα δεν ε, έχει πολύ ανεπτυγμένο κλάδο ε, των επιστημών του διαστήματος. Παρόλο που θέλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάρκεια της Προεδρίας και να προωθήσει το διάστημα. Τι δράσει θα προτείνετε ώστε οι πολίτες να αξιοποιήσουν ε, την πολιτική του διαστήματος για να εξυπηρετήσουμε την ευρωπαϊκή κοινωνία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ κύριο Στοσενόφσκι από τους ε, συντηρητικούς μεταρρυθμιστές, ECR. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δυνατότητα που έχουμε να συναντήσουμε τους Μαλταίους Υπουργούς κατά την έναρξη της ε, Προεδρίας τους. Πιστεύω ότι η Προεδρία σας θα είναι ε, εξαιρετική γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πολλές νομοθετικές προτάσεις ε, με τις οποίες θα ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι θα έχουμε ευκαιρία για πιο τακτικές επαφές. Πολύ πιο τακτικές και συχνές από ό,τι με προηγούμενες προεδρίες. Σε ό,τι αφορά το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα, ε, τα θέματα των τελών περιαγωγής, ε, της χορήγησης συχνοτήτων στο φάσμα, ε, έχουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις λοιπόν για τη Μαλτέζικη Προεδρία στο επόμενο εξάμεινο. Πιστεύω ότι τα θέματα περιαγωγής ε, θα διευθετηθούν χάρη σε στενή συνεργασία και με τους ε, συναδέλφους σας. Ένα θέμα που έχει απομείνει κρεμές είναι τα κενά που υπάρχουν στις, ε, στα τέλη για τη μεταφορά δεδομένων, για τη μεταβίβαση δεδομένων. Ελπίζω το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία και για το θέμα αυτό. Έχουμε απόλυτη επίγνωση της δυσκολία του θέματος και της περιπλοκότητα, αλλά ελπίζουμε ότι θα σημειώσουμε όσο πρόοδο γίνεται. Επίση, ε, θα ήθελα ε, για το διάστημα να σας πω ότι φέτος θα τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα Γαλιλαίο το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Και σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την Προεδρία σας και από τα πόσα το προβάλλετε στο ευρύ κοινό. Γιατί μας έχει κοστίσει τις Παναγιά στα μάτια αυτό το πρόγραμμα Γαλιλαίο, αλλά θέλουμε να φέρει κάτι καινούριο στην καθημερινότητά μας. Είναι με, το πανηρό το πρόγραμμα, αλλά υλοποιήθηκε χάρη στη στενή συνεργασία των κρατών μελών. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο απαιτητικό και φιλόδοξο πρόγραμμα που έχετε και σε πολύ χαλεπούς καιρούς, γιατί γνωρίζουμε ότι λαμβάνετε την Προεδρία σε μια δύσκολη εποχή. είναι εκ των... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ από πλευρά των φιλελευθέρων του Υπουργού τη Μάλτα για την παρουσίασή του. Είναι τεράστιο θέμα που έχουμε ενώπιον μα η ψηφιακή ενιαία ώρα. Μα απασχολεί και η έρευνα έχει πολλά να κάνει. Η Μάλτα είναι μικρή χώρα και ένα εξάμεινο είναι μικρό χρονικό διάστημα για να τα επιτύχουν όλα. Υπάρχει ένα θέμα που υπέθετο ότι θα το παρουσιάσατε, αλλά δεν το είπατε, το παραλείψατε. Είστε υπεύθυνοι και για το ναυτιλιακό τομέα και δεν είπατε πολλά γι' αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε τι στόχου ε, θέλετε να θέσετε στον τομέα τη ναυτιλία. Είναι ένα τομέα ε, τον οποίο παρακολουθώ σε διάφορε επιτροπέ και παράλληλα. Προ τον κύριο Άτζιου, μιλήσατε για την έρευνα, την καινοτομία και για το διάστημα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, σαφές, αλλά εργάζομαι με τον ε, επίτροπό σας, ε, τον κύριο Καμίλο Βέλα, στενά. Αναφέρεται πολύ ιδιαίτερα συνεργασία μας στην ε, μπλε ανάπτυξη, στην διακυβέρνηση των ωκεανών και πολλοί πόροι πηγαίνουν σε αυτές τις προσπάθειες. Ξέρετε ότι δεν ξέρουμε πολλά για το διάστημα, αλλά ξέρουμε ακόμη λιγότερα για τους ωκεανούς. Και ξέρω ότι για τη Μάλτα είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα. Το έχουμε ακούσει και σε άλλες επιτροπές. Διότι χρειάζεται περισσότερη γνώση για τους ωκεανούς στο μέλλον η ανθρωπότης. Πείτε μου παρακαλώ για την έρευνα, όχι μόνο για το διάστημα όπως είπατε, αλλά και για τους ωκεανούς τι προτεραιότητες έχετε τόσο ώστε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητε που έχουμε σε Ευρώπη. Γιατί η Μάλτα είναι πραγματικά, ε, περιβρέχεται τριγύρω από θάλασσα η κυρία Σακοράφα, που είναι η συγκίτριά μας για το πρίμα, όχι μόνο εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω την ικανοποίησή μου σαν εισηγήτρια που η Μαλτέζικη Προεδρία έθεσε σαν πρώτη της προτεραιότητα ε, την ε, ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση πρίμα στα οπλέσια του, και στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας μια από τις σπάνιες προσπάθειες επιστημονικής διπλωματίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αναγκαστικού εκπατρισμού των κατοίκων της Μεσογείου, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να προωθήσει στους τομείς των συστημάτων γεωρικών προϊόντων και διατροφής και της διαχείρισης του νερού, μια πληρέστερη ενσωμάτωση σε επιστημονικό, διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο των χωρών και, από τις δύο πλευρές της ε, Μεσογείου. Κύριε Γραμματέα, με δεδομένη την ανάγκη για την έγκαιρη έναρξη της υλοποίησης του πρίμα από μία πρώτου του 2018, όπως είπα και το πρωί στην Επιτροπή, προσβλέπω στη δημιουργική συνεργασία Συμβουλίου Επιτροπής και Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας διαβεβαιώνω σαν εισηγήτρια ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα, σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στο έργο σας ως προεδρεύοντες αυτό το εξάμεινο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σακοράφα. Η κυρία Κάπελ, εξ ονόματος του ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ. Η παρουσία σας ε, έχει πολλά καθήκοντα για την ψηφιοποίηση. Δηλαδή την ε, εισαγωγή της Ευρώπης στην κοινωνία των Gigabyte. Είπατε ότι η ψηφιοποίηση θεωρείται ότι είναι μια βασική προτεραιότητά σας και ιδιαίτερη αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα για την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Και νομίζω ότι είναι πολλά θέματα που ενδιαφέρουν και το σώμα μας που έχει να κάνει με το σύστημα των τηλεπικοινωνιών πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα το Wi-Fi για την Ευρώπη, Χθε κάναμε μια συζήτηση γι' αυτό, όπου το σημαντικό είναι να υπάρχει δωρεάν ίντερνετ για όλους τους πολίτες της Ευρώπης και ιδιαίτερα βεβαίως ε, να υπάρχει δυνατότητα να παίξει ρόλο και στον τομέα της υγείας και προβλέπονται 120 εκατομμύρια ε, ε, ευρώ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εκατομμύρια σημείων Wi-Fi και η χρηματοδότηση θα γίνει και από τα κράτη-μέλη. Ερώτηση λοιπόν, θα κάνετε ό,τι μπορείτε ούτως ώστε τα κράτη-μέλη έγκαιρα να διαθέσουν τους πόρους ούτω ώστε να εφαρμοστεί το Wi-Fi για την Ευρώπη. Άλλη ερώτηση. Το σχέδιο δράσης για τα 5G. Και εδώ επίκειται πρωτοβουλία. Το 5G είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και για να έχουμε ηγετικό ρόλο στην τεχνολογία παγκόσμια και να διατηρήσουμε αυτό το ρόλο. Η τεχνολογία 5G θα πρέπει να ξεκινήσει το 2020 και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν τεστ μέχρι το 2018 για να έχουμε τις παγκόσμιες προδιαγραφές και τα κράτη-μέλη μέχρι το 2018 θα πρέπει να υποβάλουν σχέδια για την υποδομή 5G στην επικράτειά τους. Τι θα κάνετε λοιπόν, έχετε προγράμματα, ούτω ώστε να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν αυτές τις δράσεις για τα 5G εγκαίρως και ταχαίως και να τα εφαρμόσουν πλήρως. Και για τον κύριο Υφυπουργό, ο ορίζον 2020 μπορεί να έχει προβλήματα εφαρμογής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ιδιαίτερα για τις τρίτες χώρες, όπου υπάρχουν πολλές γραφειοκρατικές δυσχέρειες. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να έχουμε μια απρόσκοπτη εφαρμογή. Και εδώ το θέμα της, χρηματο... χρηματοδότησης. 200 εκατομμύρια πρέπει να προκύψουν από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Πώς θα δώσετε τα αναγκαία κίνητρα στα κράτη-μέλη να δώσουν αυτά τα χρήματα και αν ε, κάποιες ε, χώρες δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα τις ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν και ο Κοπέρνικος πέρα από το Γαλιλαίο είναι μια δεύτερη εμβληματική προτεραιότητα στο διάστημα. Θα ε, εκτοξεύσουμε έναν δορυφόρο φέτος. Θα χρειαστούμε ως περισσότερους σπόρους. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί επαρκώς ο Κοπέρνικος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όλες τις ερωτήσεις θέσατε αφού έληξε ο χρόνος που είχατε στη διάθεσή σας, αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρούμπικ τώρα. Äh, Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον δόκτορα Μαλιά που είπε πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή αγορά και ο στόχος μας είναι να υπάρξει γνήσια ψηφιακή αγορά όπου ο ανταγωνισμός να είναι τεχνολογικά ουδέτερος μεταξύ, το... μεταξύ των υπηρεσιών Wi-Fi και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και να έχουν τις καλύτερες προσφορές οι πολίτες με σωστό ανταγωνισμό. Πολλά έχουμε κάνει για την κατάργηση του τέλους περιαγωγής, τουλάχιστον ε, να μπορούν ε, να έχουν σωστό ανταγωνισμό οι εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών, αλλά δεν υπάρχει διεθνή ανταγωνισμό. Ο στόχο μέχρι το 2019 είναι να ανοίξουν αγορέ στο εσωτερικό τη Ευρώπη. Ούτω ώστε να γίνει πραγματικότητα η ψηφιακή ενιαία αγορά. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η τιμή ε, της κατανάλωσης ε, ίντερνετ είναι 277 για κάθε γιγαμπάιτ. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε την τιμή. Αυτό θα με ενδιαφέρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγια. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω με τη σειρά μου τη Μαλτέζικη Προεδρία και να διαβεβαιώσω τους Υπουργούς ότι σίγουρα θα υπάρχει χώρος ε, συνεργασίας. Πιστεύω ότι αυτή η Προεδρία ξεκινά σε μια περίοδο που ε, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Κάποια πράγματα έχουν ολοκληρωθεί και κάποια άλλα, χάρη στη δουλειά σας, θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν γρήγορα. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η περίοδος. Κάποιες μικρές αναφορές όσον αφορά κάποια πράγματα τα οποία έχουν κρυφεί ήδη, αλλά πρέπει να υπάρχει και παρουσία του Συμβουλού για να ε, ξεκινήσει η εφαρμογή τους. Παραδείγματος χάρη, εγώ ήμουν εισηγήτρια της διάταξης ε, για την απελευθέρωση των ε, συχνοτήτων ε, πάνω από τα 700 MHz που θα ψηφίσουμε ε, αύριο στην Επιτροπή μας. Ε, θα πρέπει όμως εσείς να κάνετε κάτι ώστε τα κράτη-μέλη να φροντίσουν αυτόνομα μεν, αλλά πολύ γρήγορα δε, να προσφέρουν δυνατότητες για να ξεκινήσει και η εφαρμογή του 5G. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει και ευρωπαϊκό συντονισμό και να προσέξει η Ευρώπη βεβαίω, γιατί αυτέ οι πολύ μεγάλε αλλαγέ τεχνολογικού χαρακτήρα ε, ορισμένες φορές μπορεί να ε, δώσουν και μια νέα όθηση στο παραγωγικό ιστό και στην παραγωγική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι λίγο πιο συντονισμένο το όραμά μας. Ε, σήμερα το πρωί συζητήσαμε και ξέρω ότι δεσμεύεται η Μαλτέζικη Προεδρία να ολοκληρώσει ε, το θέμα αυτό. Ε, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και τις ε, χρηματοοικονομικές πτυχές. Όλες οι οικονομικές πτυχές πολύ συχνά μας ανησυχούν. Ε, και επίσης πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, διότι και εσείς προωθήσατε αυτή την επιλογή, διότι μία εταιρική σχέση βάσει του άρθρου 185, όπως προβλέπετε για το πρίμα, είναι πάρα πολύ δεσμευτική. Και επομένω ε, θα πρέπει να υπάρχουν και όλα όσα προβλέπονται από αυτή την πλατφόρμα. Γιατί αλλιώ ε, θα χάσουμε το στόχο που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Έχουμε καθήκον και ενώπιον των χωρών ε, με τι οποίε συνάψαμε αυτή την εταιρική σχέση να του δείξουμε ότι η γραφειοκρατία, οι περίπλοκε διαδικασίε μα μπορεί να λειτουργήσουν. Γιατί αυτέ οι πρωτοβουλίε, όπω είπατε και εσεί, είναι πολύ σημαντικέ για την εξέλιξη των αφρικανικών χωρών αλλά και τι υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει απέναντί του closing the list of our speakers. thank you very much. Η τελευταία μιλήτρια, η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Ε, δεν θα μακρηγορήσω. Εύχομαι καλή επιτυχία στη Μαλτέζικη Προεδρία και προσβλέπω σε στενή συνεργασία. Και μάλιστα ε, πρώτο θέμα τριμερούς διαλόγου ήταν η δική μου έκθεση για, το, για την περιαγωγή. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ε, και μάλιστα είχαμε συναντηθεί με τον Υπουργό Μαλέγια πριν τα Χριστούγεννα για να ετοιμαστούμε για αυτή τη συζήτηση. Και όπως είπε ο κύριος Στοσενόφσκι, περιμένουμε την ψηφιακή επανάσταση στη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας. Πολύ ενδιαφέροντας καιροί και πραγματικά ε, είμαστε προσανατολισμένοι προς το μέλλον. Επίσης, ε, ετοιμαζόμαστε και για το πακέτο της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά και οι μαλτέζικες προτεραιότητες για την ενέργεια είναι πολύ σημαντικές. Ε, ενεργειακή ανακαίνιση των κτηρίων για να γίνουν πιο αποδοτικά. Όλα αυτά μας ενδιαφέρει. Θα πρέπει να δουν και οι πολίτες πώς μπορεί να τους βοηθήσει η Ευρώπη για να ξεφύγουν από την ενεργειακή και να προσαρμόσουν τα κτίρια τους στις δυνατότητες που δίνει το μέλλον. Είτε μένουν στον ψυχρό βορρά είτε στον ηλιόλου στον νότο. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που θα έχουμε και την προθυμία σας να συντονίσετε τα μέλη του Συμβουλίου. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη συζητήσει, γιατί υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα, αλλά για μας προέχει το συμφέρον των καταναλωτών, των χρηστών, των δεδομένων, των συμπολιτών μας. Γιατί το θέμα των δεδομένων δεν έχει μόνο οικονομική πτυχή, εδώ δημιουργούμε ολόκληρη ψηφιακή οικονομία. Ευχαριστώ και περνάμε σε απαντήσεις. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Υπουργό Μαλέγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα ενθαρρυντικά σας ε, λόγια, για την εμψύχωση που μας δώσατε και για την προθυμία σας για στενή συνεργασία. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και να σχολιάσω τις παρατηρήσεις σας. Η κυρία Καρστίγιο έκανε μια σύντομη αναφορά των περισσότερων θεμάτων και σε ό,τι αφορά τον κώδικα τηλεπικοινωνιών θα ήθελα να πω ότι τώρα ε, φτάνουμε στην ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς και θα γίνει αυτή με αποκορύφωμα τον κώδικα τηλεοπικοινωνιών που έχει κέρια σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι βασική προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Και έχουμε πρόθεση να εφαρμόσουμε τις υποσχέσεις μας. Και η διεκπαιρέωση του κώδικα έχει μεγάλη σημασία και για μας και για την Προεδρία μας και για το Συμβούλιο. Και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει ήδη τις εργασίες και τη συζήτηση για το θέμα αυτό ε, με μία κατάρθρον εξέταση του κώδικα. Πιστεύουμε ότι έτσι θα κάνουμε μία εξέταση του συνόλου των άρθρων του κώδικα για να διαμορφώσουμε μία σφαιρική εικόνα, να δούμε πού έγινε οι δυσκολίες και έτσι να διευκολύνουμε το έργο και των ε, επόμενων Προεδριών. Σε ό,τι αφορά την περιαγωγή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές για την πολύ επικοδομητική τους ε, ε, συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και όπως ξέρετε έχουμε τη διορία της 15ης Ιουνίου και γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, περιμένουν τουλάχιστον, προσδοκούν την κατάργηση των τελών περιαγωγής από στις 16 Ιουνίου και μετά. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε αυτή την προθεσμία και να μην διαψεύσουμε τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Και είμαι βέβαιος ότι με εργότη προσπάθεια και με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την προεργασία που έγινε στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, αλλά και στους τριμερείς διαλόγους, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση και λύση, παρά τη διάσταση απόψεων που υπάρχει για κάποια στοιχεία, για κάποια επιμέρους της πρότασης και κυρίως για το data caps. Σε ό,τι αφορά το θέμα Wi-Fi for Europe, βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο γύρω στον Απρίλιο για το θέμα του Wi-Fi. Ήδη έχουν ξεκινήσει επικοδομητικές συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο με τον αρμόδιο συγκητή και ευελπιστούμε ότι θα διεκπαιρεώσουμε αισίως αυτό το θέμα, που είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Αναφέρθηκε άλλωστε και από πολλούς ευρωβουλευτές. Ελπίζω να σας κάλυψα με τις απαντήσεις μου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ερωτήσεις της κυρίας Νταλή, θα ήθελα να πω ότι ναι, αναγνωρίζουμε ότι το φάσμα είναι περιορισμένο και ε, είναι εθνική αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή η διαχείρισή του. Βλέπω ότι η Επιτροπή σας θέλει πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του φάσματος. Καλύτερη χρήση, καλύτερο συντονισμό και διαπιστώνουμε στην πράξη ότι Κάποιες, χρήσεις, ε, κάποιες προτάσεις αφορούν τη χρήση του φάσματος στα πλαίσια της ενιαίας ψηφιακής αγοράς που θα διευκολύνουν την ε, χρήση του, των νέων διαθέσιμων συχνοτήτων. Επίσης, ε, στο τελευταίο Συμβούλιο διαπιστώσαμε κάποια διάσταση απόψεων. Πάντως, εμείς ως Προεδρία θα ενεργήσουμε ως έντιμος διαμεσολαβητής και θα προσπαθήσουμε να συντονίσουμε μια επικοδομητική συζήτηση για να σημειώσουμε πρόοδο και στο θέμα του φάσματος και της κατανομής των συχνοτήτων. Κύριε Τοσενόφσκι, είχατε χαρά να σας συναντήσω και προηγουμένως τον Δεκέμβριο Και όπως σωστά διαπιστώσατε, η Μαλτέζικη Προεδρία είναι μια ψηφιακή Προεδρία. Συμφωνώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα και μάλιστα εμπρόθεσμα, χωρίς να ξεπερνάμε τις προθεσμίες μας. Αναφερθήκατε και στο ΠΕΡΕΚ, τον αρμόδιο φορέα συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών. Υπάρχουν κάποιες ε, παράγραφοι του κώδικα που αφορούν τον ΠΕΡΕΚ. Αλλά σκεφτήκαμε ότι καλύτερα να κάνουμε μια διεξοδική ανάλυση του κώδικα και εξέταση κατά άρθρο και κατά τμήμα και μετά να περάσουμε στον κανονισμό για τον ΠΕΡΕΚ. Νομίζω ότι αυτός, αυτή είναι η καλύτερη μεθοδολογία, γιατί και ο κώδικας έχει κάποια άρθρα για τον φορέα αυτό συνεργασία των αριθμιστικών αρχών των ΜΠΕΡΕΚ. Κυρία Βιέρνικ, πώς λέγεστε, δεν ξέρω αν το προφέρω καλά το όνομά σας. Σας ζητώ συγγνώμη. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό κλάδο, την αυτιλία. Όντως, ε, στο δικό μου Υπουργείο εμπίπτει η ναυτιλία και όπως ε, σωστά είπατε, θα οργανώσουμε τον Απρίλιο ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Σωστά το επισημάνατε και έχουμε τον κύριο Τζο Μπούτς, έναν πρώην επίτροπο που ήταν ο προτεργάτης μιας ολοκληρωμένης ναυτιλιακής πολιτικής. Ο νυν επίτροπος ασχολείται με την διαχείριση των ωκεανών και αυτό την ξεκίνησε. Πολύ σημαντικό το θέμα, συμφωνώ μαζί σας. Και πέραν τούτου συζητούμε και επανεξετάζουμε το πρόγραμμα αυτής της συνάντησης που θα γίνει στις 20 Απριλίου στη Μάλτα και θα ασχοληθούμε με την διακυβέρνηση των ωκεανών, με το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και για τις γειτονικέ μας χώρες, αλλά και για πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Κάπελ. Αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Πάντως πιστεύω ότι θα προλάβουμε έγκαιρα να το ολοκληρώσουμε και σε ό,τι αφορά την πρόταση για, το 5G πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν οι προτάσεις κυρία Στόγια και ο κώδικας είναι η καλύτερη πρωτοβουλία για να υλοποιήσουμε το 5G. Κύριε Τόγια, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. και τα ευγενικά σας και θαρρυντικά σας λόγια. Οι διαπραγματεύσεις για, τα 500, για τη συχνότητα των 500 MHz θα αποτελέσει υπόδειγμα αγαστής συνεργασίας μεταξύ των κοινωτικών θεσμικών οργάνων. Τα καταφέραμε σε αυτό και ευελπιστούμε ότι τέτοια θετική συνεργασία θα έχουμε και σε άλλους κλάδους. Κύριε Ρούμπιχ. Το θέμα των τιμών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το θέμα αυτό στην Κορεπέρ και στους τριμερείς διαλόγους. Πρόημο λοιπόν να το σχολιάσω για να μην προεξοφλήσω την έκβαση των διαπραγματεύσεων που επαναλαμβάνω συνεχίζονται. Αυτά και ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας και να κάλυψα τα σχόλιά σας. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Κυρία Κούμπουλανάτρη, ευχαριστώ που, που δείχνετε κατανόηση για τη λεπτή ισορροπία που αναζητούμε στο Συμβούλιο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι έχουμε κοινούς στόχους όλοι αυτά. Και τώρα πραγματικά ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και τον ε, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε κι εσείς. Ευχαριστώ κύριε Μπούζε Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τα ενθαρρυντικά τους λόγια, για την επιτυχία της ε, θα απαντήσω και θα σχολιάσω ερωτήσεις που αφορούν την έρευνα, τη γενοτομία και το διάστημα. Θα ξεκινήσω από την ερώτηση της κυρίας Σακοράφα για το πρίμα. Όπως γνωρίζετε, το πρίμα είναι μία από τις προτεραιότητές μας ο τομέας της έρευνας και της καινοτομία, ε, ξεκινάει από το 2012 στη Βακελώνα. Συμφωνήθηκε ότι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας ήταν ε, μια ε, πρόταση του άρθρου 185. Είναι η πρώτη τέτοια προσπάθεια στην περιοχή της Μεσογείου για να έχουμε βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και της παραγωγής τροφίμων. Να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις ρίζες της μετανάστευσης και να αντιμετωπίσουμε και κάποιε από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να υπάρχουν πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου. Θέλουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο και οι λομοθετικές συζητήσεις για το πρίμα ε, στη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, θα προχωρήσουν, ελπίζουμε. Είναι πιεσμένο το χρονοδιάγραμμα, αλλά προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εγκριθεί σύντομα το πρίμα το Μάιο, ώστε ο προπολογισμό του ορίζοντα 2020 που προβλέπεται για το πρίμα να μην ε, χαθεί. Όσον αφορά την ερώτηση ε, του κύριου Αισνερ, έχουμε μία εκδήλωση Blue Med που είναι ανοιχτή στις χώρες της Μεσογείου και η Blue Med έχει επίσης και προεξάρχονται ρόλο στη διάσκεψη το Μάιο ε, η οποία θα οδηγήσει και στη δήλωση της Βαλέτα. Ερώτηση της κυρίας Καπέλ τώρα για τον ορίζοντα 2020 ε, και την κατάλληλη συμμετοχή στον ορίζοντα 2020 των τρίτων χωρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, στην ε, επικείμενη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να δούμε και το θέμα αυτό. Για το διάστημα τώρα. καλύτερα θα την, μπορούσε να την απαντήσει αυτή την ερώτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 12 δι από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα δοθούν για ε, διαστημικά προγράμματα ε, στο διάστημα 2014-2020. Είναι ουσιαστικό το ποσό αυτό και συμφωνώ ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και επιστροφή της επένδυσή μας. Ε, το πρόγραμμα της Ευρώπης σκοπεύει να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα με διάφορα μέτρα και να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια με πιο στρατηγικό τρόπο για να υποστηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι τεχνολογίες ε, του διαστήματος και η πληροφορική θα υποστηρίξουν βασικές προτεραιότητες όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση των αερίων του θερμοκηπίου, να διασφαλίσουμε ασφαλή σύνορα και να βοηθήσουμε και την ψηφιακή οικονομία μας. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για την εφαρμογή της στρατηγικής διαστήματος. Τέλος, Είμαι βέβαιος ότι το συνολικό και φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας μας στον τομέα του διαστήματος αποδεικνύει ότι προσδίδουμε στον τομέα αυτό την προτεραιότητα που του αρμόζει. Οι δυνατότητες της Μάλτας βέβαια σε θέματα διαστήματος είναι ακόμα ε, σε πολύ πρώιμο στάδιο, όπως είπε η Μίρια Μτάλη, αλλά ε, πάντα θέλουμε να προωθήσουμε κατάλληλες πρωτοβουλίες το 2017 ε, λογικά θα είναι συναρπαστικό έτος για τη Μάλτα σε θέματα διαστήματος. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το διάστημα σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό παραβάλλον, το Explora, που περιλαμβάνει ένα πλανητάριο και ένα ε, μόνιμο χώρο εκθέσεων. Σκοπεύουμε επίσης να οργανώσουμε ε, μία εκδήλωση ενημέρωσης και κατάρτισης για το Κοπέρνικους και μία ενημερωτική ε, συνεδρία στον Ιούνιο του 2017. Επίσης, η κυβέρνησή μου θα ξεκινήσει την πρώτη εθνική πολιτική διαστήματος της Μάλτας ε, που θα αντανακλά το διάστημα για την Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Θέλουμε επίσης να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρει το διάστημα. Υπάρχουν και διμερείς συζητήσεις εν εξελίξη για να βρούμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν να δημιουργήσουμε κατάλληλες δυνατότητες. Όλα αυτά σε πλήρη συνέργεια με τι συνολικέ προσπάθειες τη κυβέρνηση, ώστε η μαλτέζικη οικονομία να είναι μια οικονομία γνώση και προστιθέμενης αξία. Ε, Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ε, ε, ε, ναυτιλιακή διάσταση του Κοπέρνικους. Θα υπάρξει και ένα εργαστήριο το Μάιο του 2017 για την ναυτιλία και ετοιμάζουμε και συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανάγκη συνέχισης των διαστημικών προγραμμάτων μεταξύ των οποίων και του Κοπέρνικους. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο υπουργούς. Σας ζήτησα να είστε σύντομοι. Ε, γιατί ε, περιμένουν και άλλοι δύο συναδελφοί σας, δύο ακόμα υπουργοί ε, στην είσοδο εδώ και 10 λεπτά περίπου. Επομένω, ήταν απαραίτητο να είστε όσο το δυνατόν πιο λακωνικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση, για το γεγονός ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και την επόμενη φορά που θα έρθετε στην Επιτροπή μας θα ε, σας υποδεχτούμε πολύ ευχαρίστως. Περιμένουμε τώρα και τους συναδέλφους σας ε, υπουργού. Uh, uh, other... Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο άλλους εκπροσώπους της κυβέρνησης της Μάλτας. I'm very sorry I kept you waiting. I'm very sorry about this. It's okay. Sorry. Uh, that we've got, uh, next... Λοιπόν, τώρα η επόμενη προσκεκλημένη μας από τη Μάλτα, από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδη για την ε, πολιτική, ε, για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες. Είναι ο κύριος Κρίς Καρδόνα, υπεύθυνο Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων. Και το άλλο θέμα, οι προτεραιότητες για την ενεργειακή πολιτική, ο κύριος Κόντραντ Μιτζέ, Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Λοιπόν, για να μην ε, χρονοτριβούμε, παρακαλώ τον Υπουργό κύριο Καρντόνα να μας κάνει την παρουσίασή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως Προεδρία είμαστε θαπεπισμένη ότι η βιομηχανία πρέπει να είναι στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως ακριβώς ε, υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλοί άλλοι φορείς που συμμετέχουν. Γιατί στον τομέα αυτό δεν υπάρχουν εκκρεμή νομοθετικά θέματα. Νομίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε το οικοσύστημα εντός του οποίου λειτουργεί η βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί και κλαδική, τομεακή πολιτική, αλλά και οριζόντια προσέγγιση. Στο παρελθόν υπήρξαν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, στο Χάλιβα και για την αμυντική βιομηχανία. Και όσο περνάει ο χρόνος, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να έχουν μια πιο πραγματιστική προέγγιση για να διατηρηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ένωσης και παράλληλα να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις που να δίδει επιχειρηματική ασφάλεια και να ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες κεφαλιακές επενδύσεις. Και θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να καλύψουν τις ελλείψεις επενδύσεων που υπάρχουν στη βιομηχανία από το 2008 το Ευρωπαϊκό Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία για να αντιστραφεί αυτή η τάση έλλειψης επενδύσεων και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, για την κυκλική οικονομία και πιο πρόσφατα την πρωτοβουλία για να ενισχυθεί περισσότερο η ενιαία αγορά. Έχουμε λάβει και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με, την, με το οικοσύστημα, για παράδειγμα την κεφαλαϊκή αγορά και την ψηφιακή ενιαία αγορά. Πριν από την Προεδρία, η Μάλτα οργάνωσε μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς για να σχεδιαστεί και να ορίσουμε το θεματολόγιο για το επόμενο εξάμεινο για τη βιομηχανία. Τμήμα του Τρίου, η Προεδρία, φυσικά θα συνεχίσει την εργασία που ανέλαβε η Προεδρία της Ολλανδίας και της Σλοβακίας και οι προτεραιότητες της Προεδρίας είναι οι εξής. Τρεις. Πρώτη, ενίσχυση τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε το λειτουργικό κόστος ε, λειτουργία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, να ανοίξουμε την πόρτα του Συμβουλίου για τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, ιδιαίτερα για τις ιδιαίτερα μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στα πλαίσια της πολιτικής για τη βιομηχανία, η Προεδρία Θεωρώ ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει τη χημική βιομηχανία. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τι μελλοντικέ προοπτικέ τη ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία. Επίση, θα εξετάσουμε την κατάσταση πραγμάτων αυτή τη τόσο ενδιαφέρουσα βιομηχανία. Η πολιτική, η, συγγνώμη, ο τομέα στήριξη το, και ο τομέα των μεταφορών, η επιμελητία των μεταφορών, δηλαδή ποια είναι τα συγκριτικά μα πλεονεκτήματα που έχουμε ω Ένωση στο εσωτερικό του τομέα τη στήριξη και βοήθεια προς τη βιομηχανία για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας λόγω και της κατάστασης στην ε, διεθνή εμπορική σκηνή, ιδιαίτερα μετά τον Brexit και τη νέα κυβέρνηση Trump και την πρωτοβουλία για να αναβαθμίσουμε το οικοσύστημα για τα start-up και την αναβάθμιση γενικά της ενιαίας αγοράς. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές καινοτόμες ιδέες και αρκετό επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη, πολλέ νέε επιχειρήσει όμω δεν τα καταφέρνουν να επιζήσουν μετά τα πρώτα κρίσιμα 3-4-5 χρόνια ή μετεγκαθίστανται σε τρίτες χώρες αντί να μένουν εδώ. Η Προεδρία μας λοιπόν είναι αποφασισμένη να τις βοηθήσει αυτές τις εταιρείε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό καινοτομίε και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που έχουν. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τις διάφορες φάσεις λειτουργία των μικρομεσαίων κατά τον κύκλο ζωή του, τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν, τι δυνατότητε που υπάρχουν, για παράδειγμα πρόσβαση σε επιθέσει χρηματοδότηση, διαχείριση πόρων, η στρατηγική του, επίση ε, λειτουργικά θέματα, το ανθρώπινο δυναμικό, την αύξηση των δεξιοτήτων που πρέπει να δημιουργήσουμε και φυσικά θα είμαι σε πλήρη επαφή με την Επιτροπή σας κατά την ε, διάρκεια των πρωτοβουλειών για, την, ε, για τις εταιρείες startup και την αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς και θα καλέσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μπούζεκ, να συμμετάσχει στην άντυπη υπουργική στις 5 και 6 Απριλίου στην Βαλέτα. Κατά την συζήτηση αυτή θα συζητηθεί η αλλαγή, θα συζητηθούν οι αλλαγές και τα προβλήματα και οι πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι startup. Τώρα έχουμε επίσης την ψηφιοποίηση του κλάδου η ψηφιοποίηση, όπω ξέρετε, εδώ και μερικέ δεκαετίε έχει αλλάξει δραματικά την παραγωγή αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, ακόμη σε έναν βαθμό, και τη λειτουργία τη δημόσια διοίκηση. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι η ψηφιοποίηση αλλάζει βαθιά όλο και περισσότερο του παραδοσιακού κλάδου και τι παραδοσιακέ υπηρεσίε. Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ε, αυτοκίνητα, για παράδειγμα, οχήματα, χημικές ουσίες, τον τρόπο με τον, με τον οποίο οι τράπεζες παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ. Στα πλαίσια αυτά, οι συναλλαγές μεταξύ κατασκευαστικού κλάδου και των ε, πελατών και των προμηθευτών έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τα αυτοκίνητα, οι ιατρικές συσκευές, οι χημικές ε, ουσίες, όλα αυτά γίνονται πιο ευφυή και πιο διασυνδεδεμένα και η Προεδρία μας θα συνεχίσει να θέτει την ψηφιοποίηση στο επίκεντρο των προσπαθειών της με πολύ προσοχή. Διάβασα το σχέδιο έκθεσης που εκπώνησε ο κύριος Μπιουτιχόφερ για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Συμμερίζουμε τις απόψεις του. Υπάρχουν παράλογες καταστάσεις. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν σύμφωνα με διάφορες μελέτες να προκαλέσουν απώλειες σε θέσεις εργασίας και επισφάλεια. Ενώ από την άλλη μεριά η Ευρώπη δεν έχει επαρκές ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και κάθε χρόνο χρειαζόμαστε 180.000 ειδικού σε θέματα πληροφορική. Γι' αυτό χρειάζεται μια στρατηγική για την ψηφιοποίηση τη βιομηχανία, που πρέπει να έχει μια ισχυρή διάσταση ανάπτυξη δεξιοτήτων. Θα ήταν προπόθεση για την επιτυχία. Θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα στην κατάρτιση, την προώθηση τη διαβίου μάθηση και να διασφαλίσουμε ότι από πολύ μικρή ηλικία, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μαθαίνουν τα παιδιά τέτοιε ψηφιακέ δεξιότητε, γιατί είναι αναγκαίε και πρέπει να είναι πολύ προωθημένε να αξιοποιούνται δηλαδή πολύ, όχι μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στον τομέα της βιοτεχνίας και των μικρομεσαίων. Επιπλέον και κατά λίγο, η Προεδρία μας βεβαίως θέλει στενή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ε, συνδιάσκεψη που θα γίνει 17 Μαρτίου για τις ε, μεταφορές βιομηχανίας και θα καλέσω τον Πρόεδρο κ. Μπούζεξ σε αυτή τη ε, διάσκεψη και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Είμαι φυσικά πρόθυμος να έρθω στη Μάλτα. 5 και 6 Απριλίου. Κανονικά συμπίπτει βέβαια με την Ολομέλεια του Στρασβούργου. 17 Μαρτίου με βολεύει καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάντως για τις προσκλήσεις. Περνάμε τώρα στην ενεργειακή πολιτική και στον Υπουργό Κόνραντ Μιτζέ. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, αγαπητοί συνάδελφοι. Νιώθω μεγάλο προνόμιο που βρίσκομαι εδώ για δύο κυρίω λόγου. Καταρχήν, το Μάρτιο 2013 συμμετείχα για πρώτη φορά στο Συμβούλιο, ε, τότε που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τα σύνδρομα που έχουμε στην ενέργεια και τι προκλήσει τεράστιε έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα γίνομαι μάρτυρα τη ε, ανάπτυξη τη ιδέα τη Ενεργειακή Ένωση. Συμμετείχα από τα σπάργανά τη στην ιδέα αυτή ε, και συμμετείχα στη διαμόρφωση της πολιτικής κατεύθυνσης ε, ως υπουργό του Συμβουλίου Υπουργών. Και τρίτον, έρχομαι σήμερα εδώ ως υπουργό από, μια, από τη μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή μάλιστα που η Ένωση αυτή προωθεί ένα πολύ φιλόδοξο ενεργειακό θεματολόγιο που θα φροντίσουμε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Κατά τύχη, μάλιστα το Μάρτιο στη θα εορτάσουμε την 60 ετία από την ίδρυση της ενιαίας αγοράς από τη συνθήκη της Ρώμης του 1957 που μάλιστα δράζεται και στην συνθήκη ΚΑΧ για τη χαλιμπουργία. και μάλιστα ε, εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία που εποφελήθηκε από την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς, που είναι επιτεύγματα της Ένωσης από την έναρξή της ε, και που από την αρχή έφερε στο επίκεντρο των συζητήσεων την ενέργεια. Σήμερα βέβαια δεν μιλούμε μόνο για τον άνθρακα και το χάλιβα, όπω οι ε, ιδρυτικέ συνθήκε, Έχουμε περάσει σε άλλη φάση στην Ενεργειακή Ένωση, που όμω εξακολουθεί να είναι σημαντική, πιο σημαντική από ποτέ. Πάντω ο κύριο Μπούζεκ ήταν από του βασικού αρχιτέκτονε αυτή τη ιδέα από τους πρωτεργάτες αυτής της ιδέας. Η ενέργεια, η ενέργεια ήταν ανέκαθεν στο επίκεντρο της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής και ε, αναμενόμενο από το 1951 ε, με τη συνθήκη ε, άνθρακα και χάλιβα. Και μάλιστα παρόλα αυτά οι κοινοτικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό είναι σχετικά καινούργια. Μόνο το 1996 είχαμε το πρώτο ενεργειακό πακέτο από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία το δεύτερο το 2003 και το τρίτο το 2009. Και μέχρι τα δεκαετία του 1990 η ενεργειακή αγορά χαρακτηρίζονταν από κρατικό μονοπόλιο και είχαμε κατακόρυφη ολοκλήρωση επιχειρήσεων σε όλες τις φάσεις ε, της παραγωγής μέχρι την πώληση. Και μάλιστα οι πρώτες οδηγίες 96 και 98 για το ηλεκτρικό ρεύμα και το αέριο προσπάθησαν να ανοίξουν την αγορά προς τον ανταγωνισμό και στη δεύτερη φάση των οδηγιών ζητήσαμε πλήρη απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών. Βέβαια, οι προσπάθειες αυτές ε, δεν ε, ευωδόθηκαν και στο... Έχουμε αρκετό έλεγχο της ε, ενεργειακής αγοράς ε, και εμποδίζουμε την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων. Έχουμε κερδίσει των τιμών. Ε, εμείς προσπαθήσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αλλάξει αυτή τη διάρθρωση της αγοράς προτείνοντας το τρίτο ε, πακέτο. Βέβαια, στο παρελθόν είχαμε αποτύχει να επιτύχουμε μια ολοκλήρωση ενεργειακής αγοράς και μάλιστα έτσι οδηγηθήκαμε και στην ε, χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τώρα όμως περνάμε σε μια νέα φάση, το τρίτο πακέτο, με πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών. Γιατί ε, εδώ και καιρό θεωρείται η ενεργειακή πολιτική ως ε, μεταβατική πολιτική. Ως πολιτική μάλλον που ήταν συνεχώ σε μετάβαση και ακόμη δεν έχουμε υλοποιήσει αυτή τη μετάβαση. Βέβαια είχαμε ε, σταδιακές διακοπές στην παροχή του αερίου και πολλά προβλήματα και η αντίρρητη πραγματικότητα μας προσγείωσε. Μάλιστα, επειδή έχουμε μία χώρα διαμετακόμισης και ε, λίγους ε, προμηθευτές, ε, κάτι που ε, μας τι ε, τις αδυναμίες μας και την ανάγκη διαφοροποίηση των προμηθευτών. Και μάλιστα, παρά την ασφάλεια αναφοδιασμού, οι ψηλές των ενεργειακών προϊόντων είναι πολύ υψηλότερε από ό,τι στην Αμερική, για παράδειγμα. Και μάλιστα, κάποια στιγμή είχαμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ τη μέρα λογαριασμό ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθούμε τις ε, ενεργειακές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, γιατί οι τιμές ενέργειας ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μισές από ό,τι οι ευρωπαϊκές. Επαναλαμβάνω, η κρίση που στο μεταξύ έλαβε χώρα μας έδωσε μια νέα όθηση ώστε να επιταχύνουμε τις εργασίες για την Ενεργειακή Ένωση και δημιουργήθηκε μια μεγάλη όθηση σε αυτό το πρόγραμμα της Ενεργειακής Ένωσης. Έτσι, με το πακέτο και τη μέτρων που έχουμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προωθήσουμε τις εργασίες ώστε στο μέλλον να μην επαναληφθούν οι αγωνίες του 2014. Θέλουμε περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών και διασυνδεσιμότητα των συστημάτων αερίου και ηλεκτρισμού. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μέσω της απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Και μάλιστα 60 χρόνια μετά την έναρξη αυτής της διαδικασίας συνεχίζουμε τις εργασίες ε, στα πλαίσια και της Μαλτέζικης ε, Προεδρίας σε αυτή την ιστορική στιγμή. Και μάλιστα η Μάλτα σκοπεύει να, να προωθήσει αυτό το θέμα στην Προεδρία της, εκπροσωπώντας 28 χώρες μέλη. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αυτό δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αντίθετα είναι ε, διαπίστωση ρεαλιστική. Και έχουμε μεγάλες διαφορές. Ε, ε, ούτε είχαμε αντιμετωπίσει τις κρίσεις κεντρικής και βόρειας Ευρώπης με το φυσικό αέριο. Και, αλλά έχουμε μια νέα κυβέρνηση που θέτει την ενέργεια ως ύψητη προτεραιότητα του προγράμματός μας. Και άσχετα με το πόσο μεγάλη είναι μια χώρα ή που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ενδιαφέρεται για την ενέργεια, γιατί η ενέργεια αφορά τους πολίτες, ε, γι' αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Και αυτό κάνουμε την τελευταία τετραετία στη Μάλτα και ξέρουμε ότι είναι τεράστιες οι προκλήσεις Θέλουμε ε, μεγάλα επίπεδα διασύνδεσης στο ρεύμα και στο αέριο και μάλιστα ακριβώς επειδή είμαστε ένα νησί έχουμε μεγάλες προκλήσεις σε ό,τι φορά την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Και ο νησιώτικος χαρακτήρας ε, φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και δίνουμε έμφαση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, δεδομένων του γεωγραφικού και φυσικού περιορισμού που αντιμετωπίζουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν ζούμε σε ένα, παρόλο που ζούμε σε ένα μικρό ε, κόσμο, δεν ε, έχουμε άγνοια για τα προβλήματα των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Και θα προωθήσουμε όλο τον ενεργειακό προβληματισμό, γιατί θέλουμε την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών, για να μην απολέσουμε και άλλε θέσει απασχόληση. Επαναλαμβάνω, η ενέργεια είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα, ε, ήταν και τη κυβέρνηση, ήταν και τη Προεδρία. Και μάλιστα η τα μεταρρυθμίσεις που έχαμε συνάδουν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Προεδρίας ε, για προσιτές τιμές, για ασφάλεια του ανεφοδιασμού ε, και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα, βιωσιμότητα, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και στι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χαμηλές τιμές στην παραγωγή ενέργειας. Έχουμε επίγνωση λοιπόν των προβλημάτων αλλά και των σημαντικών προκλήσεων. Γι' αυτό και διαβεβαίωσα και το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υποστηρίξουμε το, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση. Είναι αυτονόητο βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να το διατρανώσω για να δείτε και από αυτή τη σκοπιά τη Μαλτέζικη Προεδρία. Την Προεδρία μιας ε, ρεαλιστικής χώρας που δεν έχει ε, κανένα παραλήρημα μεγαλείου, αλλά ε, χαρακτηρίζεται κυρίως από ρεαλισμό. Και πριν περάσουμε στη συζήτηση για κανονισμούς, οδηγίες και τριμερείς διαλόγους και άλλες διαδικασίες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να παραμείνουμε ρεαλιστές και να καταλάβουμε την πραγματικότητα στην οποία ζουν οι πολίτες μας, γιατί ενέργεια σημαίνει ανάγκες των πολιτών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ε, τις ανάγκες των πολιτών, την αναζήτηση της ταυτότητάς τους και να επαναφέρουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο κοντά στους πολίτες. Έτσι θα απαντήσουμε στον προβληματισμό τους, ε, γιατί φυσικά ο κόσμος δεν μιλάει για διασυνδέσεις ε, και για αγωγούς, αλλά μιλούν ε, για τις διακοπές ρεύματο, για τους υψηλούς λογαριασμούς του ρεύματο, για το πώς θα θερμάνουν τις κατοικίες τους. Αυτά τους απασχολούν. Για πολλά χρόνια μιλούσαμε για την αθαλομίχλη για τα αιωρούμενα σωματίδια και γι' αυτό ζητήσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να βελτιώσουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση. Και θέλω όταν μας βλέπει ο κόσμος στη τηλεοράση τους να βλέπουν ότι δεν κοφεύουμε στις ανάγκες τους και στις προσδοκίες τους, αλλά αφογκραζόμαστε τις επιθυμίες τους. Και αυτό ισχύει περισσότερο για την ενέργεια που βρίσκεται στο επίκεντρο των, α, του ευρωπαϊκού προβληματισμού. Μόνο έτσι θα έχουμε μια αμοιβαίως επωφελή κατάσταση και για τις πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν αφογκραστούμε τον προβληματισμό των απλών πολιτών, τότε κάποιο άλλο θα το κάνει. Σημαντικέ οι προκλήσει λοιπόν και τη Προεδρία και των θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστέ και πραγματιστέ, προσφέροντα απτέ λύσει σε ουσιαστικά προβλήματα. Θεωρώ ότι το πακέτο Ενέργεια για όλου του πολίτε μπορεί να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσει την καθημερινότητα. Και μαζί με τον ε, ε, Μάρο Σεύσοβιτς ε, και τον, και τον Επίτροπο Αρίας Κανιέτε θα συνεργαστούμε ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτό το σχέδιο. Θέλουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των πολιτών, στις ανησυχίες τους και καλύτερη και πιο κατάλληλη για το ρόλο αυτό είναι οι ευρωβουλευτές που έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες. Και γι' αυτό η Προεδρία μας χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο από ποτέ. Αν θέλουμε να, να προσανατολίσουμε το Συμβούλιο στις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Εμείς θα ακολουθήσουμε τις βασικές μας προτεραιότητες. Καταρχήν, ε, πρόταση για το Gas ε, SOS, την εξασφάλιση αναφοδιασμού του αερίου. Επίσης, ε, ενέργεια, καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους και δημιουργία ε, όθηση στο νέο πακέτο και σημαντικό ε, θέμα η ευρωμεσογειακή διάσταση. Ό,τι αφορά τον αναφοδιασμό σε φυσικό αέριο, είναι ακρογωνία λήθο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προτεραιότητα τη Μαλτέζικη Προεδρία. Και γι' αυτό θέλουμε να επικεντρωθούμε ε, στο θέμα αυτό. Ήδη είχαμε αρκετέ επαφέ και συνεδριάσει ακολουθώντας την όθηση της Σλοβακικής Προεδρίας. Θα συνεχίσουμε τις, προσπάθειες αυτές και των προηγούμενων Προεδριών και ελπίζω ότι το Συμβούλιο σύντομα θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ασφάλεια των εφοδιασμών σε φυσικό αέριο. Ελπίζω ότι θα είναι αγαστή συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για, τον, ε, για την ασφάλεια του ε, ενεργειακού ανεφοδιασμού και ελπίζω να καταλήξουμε στη συμφωνία πριν το τέλος της ε, Μαλτέζικης Προεδρίας. Ε, Επίση αποδίδουμε ιδιαίτερη προσπάθεια στα επιμέρους στοιχεία αυτού του θέματο. Περιφερειακή συνεργασία, για παράδειγμα. Σημαντικό θέμα, η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με βάση ομάδες ε, ε, κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην προμήθειά τους σε φυσικό αέριο. Επίση, θα ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Σημαντικό θέμα για την ασφάλεια του ανεμφοδιασμού. Και φυσικά θα πρέπει να κρατήσουμε ε, χαμηλή τη γραφειοκρατία και προσπίζοντας την εμπιστευτικότητα τέτοιων πληροφοριών. Και τα ε, συμβόλαια αυτά για, τα, για την προμήθεια, που είναι το 40% ε, των ενεργειακών συμβολέων, θα πρέπει να διακυβεύσουν την ασφάλεια αυτή του ανεφοδιασμού. Επίσης, ό,τι αφορά τις συμβάσεις για το αέριο, και δεν πληρούν το κατόφλι το 40%, οι αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ζητούν και άλλες πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια των εφοδιασμού. Βέβαια, αρκεί να μην περιλαμβάνει τιμές και να λαμβάνει υπόψη ε, το ανάλογο ε, γραφειοκρατικό ε, κόστος. Τώρα, αλληλεγγύη. Θα πρέπει να είναι η ίστατη λύση, αφού έχουν εξαντληθεί, έχουν όλα τα προηγούμενα μέτρα. Επίσης, η ελεγγύη μαζί με τις πιθανές αντισταθμίσεις θα είναι το τελευταίο σκέλος του κανονισμού. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Και προσβλέπω σε στενή συνεργασία ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άμεση πρόοδο, για να ε, βελτιώσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Ελπίζουμε να υπάρχει συνεργασία και να προχωρήσουμε με το Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν ε, ε, εντομότερα. Περνάω τώρα στο θέμα της επισήμενσης για την ενέργεια. Αυτός είναι ένας από τους ε, τομείς τους οποίους θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα για τη Μαλτέζικη Προεδρία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερήσουμε κι άλλο για κάποια πράγματα τα οποία εκκρεμούν εδώ και καιρό. Πρέπει να προχωρήσουμε για να επικεντρωθούμε στην καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους. Με αυτό κατά νου η Μαλτέζικη Προεδρία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέβρεση λύσει. Ε, επικροτούμε τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και ε, πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πρόοδο. Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τώρα περνάω στις προθέσεις μας για την δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια για όλους. Η Ευρώπη δεσμεύεται να δημιουργήσει μια ενεργειακή ένωση βάσει την ενεργειακή ε, πολιτική και το πλαίσιο που συζητήθηκε το 2014 για την πολιτική για το 2030. Εγκρίθηκαν ε, από το Σώμα των Επιτρόπων αυτές οι, ε, αυτά τα μέτρα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν την καθαρή ενέργεια για την Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσουμε βέβαια την Ενεργειακή Ένωση αλλά πρέπει να ανοίξουν και τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν μπορούμε απλώς να το δηλώνουμε. Επομένως, ε, η Ευρω... Μαλτέζικη Προεδρία θα προχωρήσει τι συζητήσει ε, και στις πέντε διακλαδώσεις, την ενεργειακή απόδοση, την σχεδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, ε, ασφάλεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διακυβέρνηση. 27 Φεβρουαρίου θα καλέσουμε τους Υπουργούς να μας πούν τις βασικές τους προτεραιότητες για αυτό το τόσο σημαντικό πακέτο. Ε, είμαστε υπέρ της αρχής της ενεργειακής απόδοσης πρώτα. Επομένως πρώτα θα εξετάσουμε την αναθεώρηση των στόχων της ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο μέχρι τα τέλη Ιουνίου για το θέμα αυτό. Έτσι θα δημιουργήσουμε και την κατάλληλη όθηση για να προωθήσουμε και τα άλλα σχέδια της ε, καθαρής ενέργειας που μόλις ανέφερα. Ε, βασιζόμαστε φυσικά και στην αγαστή συνεργασία μαζί σας για να προχωρήσουμε την πρωτοβουλία της Ενεργειακής Ένωσης στο το συντομότερο δυνατόν. Σε επίπεδο ομάδων εργασία θα αυξήσουμε και τον αριθμό των συνεδριάσεων. Ε, κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ε, προσβλέπουμε στην ανακοίνωση τη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση τη ε, Ενεργειακή Ένωση και κυρίω ε, θα επικεντρωθούμε στην περιφερειακή προσέγγιση. Ε, θέλουμε να υποστηρίξετε και την Ενεργειακή Ένωση όπως κάνατε το Νοέμβριο και ε, ενδιαφέρεστε και για την κατάλληλη πλατφόρμα. Στην τελευταία ε, συνεδρίαση ε, που ε, έγινε, που είναι και η τελευταία ε, που έγινε στη διάρκεια της Επιτροπής Βιούνκερ και του Κοινοβουλίου ε, πριν από τις διακοπές. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να προχωρήσουμε αυτή τη διάσταση. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις και μετά από το άτυπο συμβούλιο το Μάιο θα γίνει μια δεύτερη διάσκεψη υψηλού επίπεδου που θα περιλαμβάνει υπουργού και υπουργού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδιαφερομένων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις πλατφόρμες για το φυσικό αέριο, την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και θα θέλουμε φυσικά να προσκαλέσουμε και εσά, κύριε Πρόεδρε και τα μέλη της Επιτροπής να συμμετέχουν σε αυτή τη ε, διάσκεψη. Επίσης εκεί θα ξεκινήσει και ένα φόρουμ ε, μικρών ε, ε, νήσων εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπεύουμε να προωθήσουμε στη διάρκεια της προεδρίας μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού, τη βιωσιμότητα και μια ενέργεια προσιτή για όλους μας τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις και τους δύο υπουργού και να πω στους συναδέλφους ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο σχεδόν, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ε, συζήτηση. Σας παρακαλώ όμως να είστε λακωνικοί όσο το δυνατόν για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Ε, καταρχάς, εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Κάσα, ο οποίος είναι και αυτός ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τη Μάλτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς τον Υπουργό Ενέργειας. Είναι ο υπουργό ο οποίο ήταν ε, υπεύθυνο και για την ιδιωτικοποίηση τη Εν Μάλτα, που είναι η επιχείρηση ηλεκτρισμού και είναι και ε, γνωστό από τα έγγραφα του Παναμά, γιατί ξέρουμε ότι έχετε μυστικέ επιχειρήσει και υποτίθεται ότι έπρεπε να καταθέσετε ένα εκατομμύριο ευρώ σε αυτέ τι επιχειρήσει μπορείτε να εξηγήσετε στην Επιτροπή από πού προέρχονται αυτά τα εκατομμύρια. Οι Μαλτέζοι πολίτες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το Κοινοβούλιο σας θέτουν αυτές τις ερωτήσεις συνεχώς. Σήμερα λοιπόν είναι η κατάλληλη ευκαιρία να μας δώσετε τις απαντήσεις που περιμένουμε εδώ και μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλη για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να καλωσορίσω τους Υπουργούς Καρντόνα και Μίτσι και θα ήθελα ως μέλος της Επιτροπής ε, να σας πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας ε, στο πρόγραμμα που μας παρουσίασετε Και επιτρέψτε μου επίσης, επίσης, γιατί και εγώ είμαι από τη Μάλτα, να πω ότι για τη χώρα μας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη συγκυρία, το γεγονός ότι έχουμε πλέον Μαλτέζικη Προεδρία. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Μίτσι. Ε, με χαρά άκουσα ότι σας ενδιαφέρει η πρόσβαση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να ξέρω σε τι θα επικεντρωθείτε περισσότερο και πώς σκοπεύετε να βοηθήσετε τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις startups. Κύριε Μίτσι, είστε διάσημος γιατί περάσατε από τα βαρέα καύσιμα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και αυτά ε, τα καύσιμα πλέον ε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο κανονισμός για την ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτού του κανονισμού είναι η ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και αν βρίσκονται, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσεων. Πώς σκέφτεται η Προεδρία να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και πού μπορεί να έχει πλειοψηφία η Προεδρία για το θέμα αυτό. Ο κύριος Τούρμες, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ασχοληθώ για τα θέματα ενέργειας και ο συνάδελφος κύριος Μπουτικόφερ θα κάνει μια άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε την Προεδρία σας για να εργαστούμε για την περιφερειακή διάσταση γύρω από τη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως έχουμε πει και εμείς στο Κοινοβούλιο Τώρα έχουμε μία επίσημη μορφή συνεργασίας για τη Βαλτική, για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης για τη Βόρεια Θάλασσα. Ε, εργαζόμεθα πολύ η Γερμανία, Γαλλία και Μπενελούξ. Έχουμε λοιπόν κάποια δραστηριότητα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την Προεδρία σας για να εμβαθύνουμε τη συνεργασία για την ενεργειακή απόδοση, τα δίκτυα, τις αγορές και τις ανανεώσιμες μεταξύ των χωρών της ε, Μεσογείου με τους εταίρους μας δηλαδή από την άλλη πλευρά. Και προσβλέπω στην ε, εργασία για το θέμα αυτό. Τώρα, όταν λέτε ότι οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλές ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις μας, πρέπει να κάνετε μια διαφοροποίηση. Για το φυσικό αέριο, ναι, σε ένα βαθμό ισχύει. Αλλά κοιτάξτε την εξέλιξη των τιμών του φυσικού αερίου. Λόγω της ενίας αγοράς και όλων των ενεργειών μας και λόγω του υγροποιημένου φυσικού αερίου και επειδή, επειδή είναι συνδεδεμένα και με τις τιμές του πετρελαίου, η, κατεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου. Τώρα είναι πολύ μικρότερη η διαφορά από την τιμή του φυσικού αερίου από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Επίσης, η χονδρική τιμή για την, για την τιμή για τη βιομηχανία ήταν 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι γύρω στα 30 στην περιοχή Γαλλία, Μπενελούξ, αν δεν υπάρξει κρίση στη Γαλλία για, την, ε, για τη θέρμανση μαζί με την... Ε, ε, μαζί με τα προβλήματα του πυρηνικού τομέα. Αν δείτε τις τιμές στην Αμερική και τις συγκρίνουμε με τη δική μας τιμή, δεν ξέρω ποια σας έδωσε αυτά τα στοιχεία, αλλά θα πρέπει να τα ξαελέγξετε. Έχουμε κάνει πολλά. Πολλά από όσα έπρεπε να κάνουμε για τα έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλικιώτης για την ΚΟΕ. Ε, θέλω να καθαρολώσω τους δύο υπουργούς, τον κύριο Καστοράκη και τον κύριο Νίζη που είναι σήμερα μαζί μας. Πρώτα-πρώτα ε, να πω για τα θέματα βιομηχανίας. Εμείς ε, χαιρετίζουμε τους στόχους που έχει θέσει η Μαρτίζικη Προεδρία για την πρόθεση της ε, επαναβιομηχανοποίησης και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια δράσης. Δυστυχώ, σύμφωνα με έρευνα, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνουν κατά τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργία του εκτιμάται το κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων χάνονται 1,7 εκατομμύρια θέσει απασχόληση. Η κατάσταση χειροτερεύει γιατί εφαρμόζονται ακόμα νεοφιλελεύθερε πολιτική σκληρή λιτότητα. Το ερώτημα που μπαίνει είναι ποια συγκεκριμένα μέτρα, ακούσαμε στην εισαγωγή τη παρέμβαση αρκετά, αλλά για να στηριχτούν αυτέ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ιδιαίτερα ποια μέτρα θα λάβετε για να ενισχυθεί το πρόγραμμα COSME για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και δεύτερο, να διευκολυνθεί πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και να οθούν κίνητρα για την ανάπτυξή, κάτι που είναι ένα ε, κενό ε, στι πολιτικέ στην Ευρώπη. Το δεύτερο που ήθελα να θέσω είναι για τι ενεργειακέ πολιτικέ. Μια βασική προτεραιότητα τη δική μα τη ομάδα είναι να διασφαλιστεί η ενέργεια ως δημόσιο αγαθό, ως κοινωνικό αγαθό, να έχουν όλοι ισότιμη και ευθυνή πρόσβαση. Γίνεται μεγάλη αναφορά για το νέο φαινόμενο της ενεργειακής στόχιας. Αυτό που θέλουμε να ακούσουμε είναι αν, υπάρχουν, αν υπάρχει ένα ε, προτάσει σκέψης για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για καταπολέμηση τη ενεργειακής στόχιας. Ακόμα, επειδή η Μάρτα έχει εμπειρία και αναφέρομαι στην ενεργειακή απομόνωση κρατών μελών και περιοχών από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το στόχο που τέθηκε μέχρι το τέλος του 2015 να αρθεί αυτή η ενεργειακή απομόνωση. Θα ήθελα να σκέψεις σας γύρω από αυτόν τον τομέα. Και τέλος, στην έκθεση τη Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ενεργειακή Ένωση αναφέρεται για τα κοιτάσματα τη Ανατολική Μεσογείου. Το πόσο είναι σημαντικά να αναπτυχθούν και ιδιαίτερα η συνεργασία στη Μεσόγειο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ενίσχυση της Ευρώπης. Θα ήθελα τις δικές σας σκέψεις γύρω από αυτήν την προοπτική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Κάπελ, για το ΙΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Καρντόνα, κύριε Υπουργέ Μίτση. Καταρχά, να απευθυνθώ στον Υπουργό κύριο Μίτση. Σήμερα το πρωί είχαμε μια συζήτηση με τον Επίτροπο Ζεύκοβιτς ιδιαίτερα για το πακέτο για την καθαρή ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο και προβλέπεται ότι μέχρι το 2020 ή καλύτερα μέχρι την εφαρμογή του πακέτου, θα, μέσω της εφαρμογής του πακέτου θα αυξήσουμε κατά 1% το ΑΕΠ και θα δημιουργήσουμε 190.000 θέσεις εργασίας γενικά. Τώρα που έχει υποβληθεί αυτό το πακέτο, θεωρούμε ότι έχουμε καταθέσει το 90% των προτάσεων για την ενεργειακή πολιτική και είπατε ότι είναι πολύ σημαντική εφαρμογή αυτού του προγράμματος και η πιο αποτελεσματική εφαρμογή του. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα. Ω Συμβούλιο θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να εφαρμοστεί σύντομα το πακέτο αυτό μέσω τριλόγων και κάτι άλλο προς τον Υπουργό κ. Καρντόνα πολύ σημαντική τομή σα, ε, μικρομεσαίε, ε, βιομηχανία. Παρουσιάσατε τι προτεραιότητέ σα, αύξηση τη αγωνιστικότητα και ανάπτυξη, μείωση του κόστου των ε, συναλλαγών και ιδιαίτερα ενίσχυση του διαλόγου με όλου του εμπλεκομένου φορεί και ιδιαίτερα τι μικρομεσαίε. Είπατε όμω ότι δεν προβλέπονται νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα θέματα για τις μικρομεσαίες και για τον τομέα της ε, βιομηχανίας. Μιλήσαμε για την κυκλική οικονομία, για την κεφαλαϊκή ένωση και την ψηφιοποίηση. Όλα αυτά σχετίζονται λοιπόν με τα θέματα αυτά. Κατά την Προεδρία σας, ε, μήπως θα είχατε πιο συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναβιομηχάνηση. Έχουμε το στόχο του 20% της επαναβιομηχάνησης για την Ευρώπη. Προβλέπετε συγκεκριμένα μέτρα που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, ίσως κατά την επόμενη, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ούτω ώστε η Ευρώπη να επιτύχει αυτόν τον στόχο ή τουλάχιστον να προσεγγίσει αυτόν τον στόχο του 20% επαναβιομηχάνηση. Σας ευχαριστούμε κυρία Κάπελ. Η κυρία Μετσόλα, επίσης από τη Μάλτα. Ευχαριστώ. Υπουργέ Μίτση, ω περήφανη Μαλτέζα πολίτη, μου φαίνεται πραγματικά σα ορεαλιστικό ότι ο μόνο Μαλτέζο υπουργό που εκτίθεται από τα ε, έγγραφα του Παναμά με κρυφές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο εμφανίζεται μπροστά μας να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Κόνραντ Μίτς λέει ότι πώς ε, αποκαλύφθηκε ότι είχε ανοίξει μια εταιρεία στον Παναμά ε, ταυτόχρονα με την ανάληψη των υπουργικών του καθηκόντων και μάλιστα έχει καταθέσει τεράστια ποσά σε αυτές τις επιχειρήσεις που δεν μπορεί να έχει νομίμως κερδίσει ως υπουργός είστε αναξιόπιστος, απόλυτα αναξιόπιστος και είναι πραγματικά υπερβολη... αυτή η παρουσίαση εδώ σήμερα είναι σουρεαλιστική. Με εκνευρίζει γιατί φαίνεται ότι θα αναγκάσετε όχι μόνο του Μαλτέζου, αλλά και το Συμβούλιο να πληρώσει το δικό σα τίμημα. Έχω ερωτήσει που μόνο εσεί μπορείτε να απαντήσετε. Με το πόθεν έσχεση που έχετε υποβάλει, πώ πρόκειται να χρηματοδοτήσετε τη σε κατάθεση ενό εκατομμυρίου δολαρίου που έχει συμφωνηθεί από του οικονομικού σα συμβούλου για να ανοίξετε λογαριασμό στο Παναμά. Επίση, φαίνεται ότι ε, θα έχετε επιπλέον ε, ε, εισόδημα από κάποιες προμήθειες. Από πού θα προέρχονται. Έχετε ανοίξει τρεις εταιρείε. Ε, ε, εσείς, ο, ο προσωπάρχης σας και μια τρίτη που αναφέρετε για το Skype. Θα πείτε επιτέλους στον κόσμο ποιοι θα είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτών των εταιριών και αυτών των εισοδημάτων. Γιατί ο κόσμος πραγματικά αξίζει μια απάντηση και εμείς το ίδιο. Ευχαριστώ κυρία Βέρνερ, είναι η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει. Μία για το θέμα βιομηχανική πολιτική και μία σε εσά κύριε Μίτσε για την ενεργειακή πολιτική. Το κοινοβούλιο μα και η δική μα επιτροπή εδώ, η Ήτρε, εδώ και χρόνια ζητάει μία συνεπή βιομηχανική πολιτική και χαίρομαι που αναφερθήκατε τόσο αναλυτικά στο θέμα αυτό και νομίζω ότι τώρα εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Εδώ, χαίρετε και τώρα που εξελέγει ο Τραμπ είναι πολύ βασικό να έχουμε μια συνεπή βιομηχανική και εμπορική πολιτική στην Ευρώπη. Λοιπόν, το ερώτημα. Πώς θα δημιουργήσουμε οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη και θέσει εργασίας και την ε, ψηφιακή μετατροπή σε τόσο δυσχερή κατάσταση. Η έκκληση του Κοινοβουλίου που είχαμε και τον περασμένο Οκτώβριο μέσω ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για μια συνεπή βιομηχανική πολιτική και όπου το ζητάνε και διάφοροι φορεί όπω οι φίλοι τη βιομηχανία, όλοι αυτοί στηρίζουν αυτό μα το αίτημα. Πώ ε, μπορεί η Προεδρία σα να προωθήσει μια ενεργή βιομηχανική πολιτική για να ζητήσετε από την Κομισιόν να κάνει κάτι. Εδώ είναι η ουσία. Η Προεδρία και το Ευρωκοινοβούλιο καλούμε να υπάρξει αυτή η βιομηχανική πολιτική, αλλά δυστυχώς δεν προκύπτει τίποτα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή πολύ λίγα. Και κάτι ακόμη, να μην ξεχάσετε την πολιτική που ήδη τόνισε το Κοινοβούλιο για συγκεκριμένους τομείς, για παράδειγμα για τον τομέα του Χάλιβα και τον τομέα των σιδηροδρόμων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσετε τα θέματα αυτά. Να μην παραμείνει μόνο λόγια σε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Κύριε Μίτσε, χάρηκα που άκουσα να λέτε ότι θα ασχοληθείτε με τόσες λεπτομέρειες και τόσο ενεργά με την ενεργειακή πολιτική, μια φράση είπατε. Η ενέργεια αφορά τους ανθρώπους, τους πολίτες. Και χαίρομαι και πολύ που αναφερθήκατε στην επισήμανση ενεργειακής απόδοσης. Για το θέμα αυτό είμαστε ακόμη κολλημένοι στον τριμερή διάλογο. Αν θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες μας ότι θέλουμε να υπάρχει ενεργή για τους πολίτες ε, ενεργειακή πολιτική, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν πραγματικά να κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτω ώστε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας επιτέλους να έχουμε επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Κόχλιτσεκ. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν πρόκειται να μακρηγορήσω όπω οι συνάδελφοι. Πριν ε, λίγα χρόνια κάποιος ε, κατασκευαστής μετρητών άνοιξε ένα, μια θηγατρική στη Μάλτα, ένα υποκατάστημα. Ε, συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε αυτό το τομέα. Επίσης, ποιος, ε, ποιο είναι το σχέδιό σας για να επιτύχετε το στόχο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προτιμάτε την αιωλική ενέργεια, τη γεωθερμική ενέργεια ή τα φωτοβολταϊκά. Φαντάζομαι θα έχετε κάποιο ποσοστό για το στόχο σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη Μάλτα. Ευχαριστώ κύριος Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό Καρντόνα. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στο θέμα της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στις δεξιότητες Σας διαβεβαιώ ότι πολύ ευχαριστώ και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλουμε στη συζήτηση και να ακούσουμε και τη γνώμη των ενδιαφερομένων φορέων της Μάλτας για το θέμα αυτό. Επίσης, ποιος είναι ο κίνδυνος από πιθανές ε, συμμετοχή τρίτων χωρών στην ε, ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Μπορούμε να προβλέψουμε κάποια συμπληρωματικά μέτρα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τον ε, κύριο Μίτσε. Πώς μπορείτε να είστε προεδρεύον στο Συμβούλιο Ενέργειας όταν έχετε χάσει αυτό το χαρτοφυλάκιο στη χώρα σας. Σας το έχουν αφαιρέσει εξαιτία τη ανάμειξή σα στο σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρίφιν. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γέζη. Υπουργέ Μίτσι, άκουσα με ιδιαίτερη χαρά να αναφέρεστε σε 28 χώρε μέλη. Ε, την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλη είπε κάποιο ότι είναι ηρωνικό η Μάλτα να είναι προεδρεύουσα όταν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο είμαστε εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το σύνολο τη Ευρώπη. Κύριε Καρντόν, άκουσα με ιδιαίτερη χαρά ότι η κατάρτιση και οι δεξιότητε ε, βρίσκονται στο επίκεντρο τη βιομηχανική σα πολιτική. Και η Υπουργέ Μίτσε, είπατε ότι η ενέργεια αφορά κυρίω του ανθρώπου. Εμεί, ω Σοσιαλιστέ και δημοκράτε, πιστεύουμε ότι η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα είναι ένα, ένα στοιχειώδες κοινωνικό δικαίωμα. Έχουμε πάνω από 50 εκατομμύρια συμπολίτες μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνθήκες ε, ενεργειακής φτώχειας. Έχουμε το μανιφέστο στην ε, πολιτική μας ομάδα για την ενέργεια και θα ε, γίνει, ε, γίνουν τα εγγένεια στην Γάνδη. Μάλιστα, εγώ ως ε, Ευρωβουλευτής από τη Βόρεια Ευρώπη είπα ότι κανείς δεν θα πρέπει στην Ευρώπη να πρέπει να κάνει μια επιλογή μεταξύ της θέρμανσης και της, ε, τροφής, διατροφής του. Η Ντάλη τότε είπε Τερέζα στις ε, μεσογειακές χώρες το καλοκαίρι έχουμε κόσμο που πεθαίνει γιατί δεν, δεν μπορεί να πληρώσει το κλιματισμό και πεθαίνουν από τον καύσωνα. Οπότε έχουμε και ένα αλλακτικό ε, σύνθημα. Κανένας δεν θα πρέπει να, πρέπει ε, δεν θα πρέπει να ε, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μεταξύ της θέρμανσης, της ψήξης ή της διατροφής. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε την ενεργειακή φτώχεια και χαίρομαι που ο μετριασμός της βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τις ερωτήσεις από τα μέλη και τώρα θα ήθελα να ζητήσω και από τους δύο υπουργούς, ίσως να ξεκινήσουμε από εσά, να απαντήσουν. Με την ίδια σειρά, αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν τον λόγο Είναι μικρό μου το, χαρτοφυλάκιο, το τμήμα του χαρτοφυλακίου μου στην Επιτροπή σας, επομένως μπορώ να απαντήσω ε, σε δύο σκέλη. Θα ξεκινήσω με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, προφανώς και η πρόσβαση ε, σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις ε, είναι ζωτική σημασία. Και έχουμε διαπιστώσει, τουλάχιστον αυτό έχω δει στα τέσσερα ε, χρόνια μου ως Υπουργός Οικονομίας ε, που συμμετέχω και στα Συμβούλια Οικονομίας, έχουμε θέσει στο θεματολόγιο πρόσβαση στη χρηματοδότηση επανειλημμένως. Έχουμε όμως διαπιστώσει επίσης ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσμα απαραίτητο. Και όπως ε, ανέφερε και ο κύριος Μπούτικόφερ όσον αφορά τη βιομηχανία, οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός ε, της Ευρωπαϊκής Επικρότητας αντιμετωπίζουν και ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Επομένως, ε, φιλοδοξία μας ως Προεδρία είναι να υπάρχει ε, κατάλληλη συζήτηση που θα προσφέρει κατάλληλες λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις νεοφυγείς επιχειρήσεις, για τις ε, ε, υπόλοιπες επιχειρήσεις για να υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα προέρχεται από ένα δάνειο από μια τράπεζα, μπορεί να είναι κίνητρα, μπορεί να είναι πρωτοβουλίες, μπορεί όλα να δοθούν υπό τη μορφή του τι κάναμε σε τοπικό επίπεδο νομοθετώντας για τις οικογενειακές οικογενειακές επιχειρήσεις, για τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις και προκειμένου να το καταφέρουμε αυτό ε, θα διοργανώσουμε ένα άτυπο συμβούλιο στο οποίο θα ασχοληθούμε με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και επίσης ε, στο επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνισμού θα έχουμε τις ε, startups και τις scale-ups, κάποιες πρωτοβουλίες για το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτές τις επιχειρήσεις και φυσικά στην Επιτροπή θα διοργανώσουμε και μια σειρά από τεχνικές συνεδριάσεις στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Από πλευρά λοιπόν μικρομεσαίων επιχειρήσεων νομίζω ότι σαφώς ε, και καταλαβαίνουμε ότι ε, πρέπει να γίνει ανταλλαγή απόψεων για την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, startups και τις scale-ups και να προσπαθήσουμε να πιέσουμε λίγο περισσότερο ε, και να βοηθήσουμε τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά ε, το βιομηχανία, και εδώ νομίζω θα μπορούσα να απαντήσω σε δύο σκέλη. Μπορώ να ξεκινήσω με τη βιομηχανική πολιτική και μετά να ολοκληρώσω με τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Το πρώτο ερώτημα που μας τίθεται είναι κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει βιομηχανική πολιτική. Αν δείτε λίγο το ιστορικό, τι συνέβη μετά από την Επιτροπή Juncker. Ε, η οποία επιτροπή αποφάσισε ότι η βιομηχανική πολιτική είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας ευρύτερη πολιτική ε, και συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Και παρά το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίε αυτές ε, αφορούν διάφορου τομεί πολιτικής, είναι όλες πρωτοβουλίε της αγορέ, που σημαίνει ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχουν και το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου ε, να έχουμε και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να βοηθήσουμε τη βιομηχανική πολιτική. Κι όμως δεν υπάρχει ακόμα βιομηχανική πολιτική. Και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής και αν υπάρξει τότε θα την προσέσουμε και στο θεματολόγιο του ε, Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Ε, για τις διάφορες αντιδράσεις, για τα όσα είπατε εδώ, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Ε, διότι ένας από τους βασικούς στόχους της Προεδρίας μας είναι να προχωρήσουμε τα όσα έκαναν οι κάτω χώρες και η Σλοβακία στη διάρκεια της δικής τους της Προεδρίας και κυρίως θα επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τρίτες χώρες. Και το κόστος ε, εργασία στην, και δραστηριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά όπως μπορείς και να δηλώσω στην εισαγωγή μου, μας ενδιαφέρει κυρίως η χημική βιομηχανία, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, ε, θέματα ε, εφοδιαστικής ε, ε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για startups και scale-ups και φυσικά το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει και επιθυμία των κρατών μελών να υπάρχει μια συνολική βιομηχανική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ως ευρύτερο θέμα συζήτησης όπως σας είπα και σκοπεύουμε να συζητήσουμε και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως κυρίο θέμα του άτυπου συμβουλίου στη Βαλέτα. Νομίζω ότι με αυτό καλύπτονται τα περισσότερα από τα όσα σχολίασαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ολοκληρώσω με την παρατήρηση της κυρίας Βέρνερ για το διακύβευμα και για το τι θα γίνει μετά από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ο πρόεδρος Τραμπ. Σαφώς και αλλάζουν τα πράγματα αλλάζουν ε, ε, τα σενάρια, αλλά κατά την άποψή μου αυτή είναι και μια καλή ευκαιρία να δράξουμε αυτή την ευκαιρία λοιπόν, να υψώσουμε τον πύχη και να βελτιώσουμε το δικό μας οικοσύστημα και να γίνει το δικό μας οικοσύστημα πιο ευνοϊκό. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι περισσότερο επιφελή σε θέματα διεθνούς εμπορίου, διεθνών οικονομικών και μπορεί να είναι και ε, μεγάλος παράγων στο διεθνές ε, σκηνικό. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και να δώσω το λόγο και σε εσά, κύριε Υπουργέ. Να αρχίσω με την ε, ερώτηση του κυρίου Τούρνε. Έθιξε πολλά πολύ σωστά θέματα. Πρώτα απ' όλα η περιφερειακή διάσταση για τη Μεσόγειο. Η Μάλτα και η Προεδρία μας θέλει να προχωρήσει, να προωθηθεί ιδιαίτερα αυτή η ευρωμεσογειακή διάσταση. Νομίζω ότι η διασυνδεσιμότητα και για θέματα ενέργειας και για άλλα θέματα τη Βόρεια Αφρική μπορεί να προσθέσει αξία για την Ευρώπη. Θα προωθήσουμε τα θέματα αυτά και ως κράτος μέλος τα έχουμε προωθήσει. Έχουμε στηρίξει την ε, αίτηση της Ιταλίας για σύνδεση με την Τινησία. Την προωθήσαμε μέσω της Κομισιόν και η Ευρωμεσογειακή Διάσταση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι κλειδί και για να έχουμε μια νοοτροπία ενεργειακής απόδοσης αλλά και για να έχουμε μια εναλλακτική πηγή ενέργειας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την ε, ασφάλεια προμήθειας. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα σταθερότητας βέβαια στη Βόρεια Αφρική. Για παράδειγμα ο γείτονάς μας η Λιβύη είναι σε κατάσταση μεγάλης αναταραχής. Είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν τέτοιες πρωτοβουλίε σε αυτή τη συγκυρία, ωστόσο θα μπορούσαμε να έρθουμε σε στενότερη επαφή με την Αλγερία, το Μαρόκο, με την Τινησία, με την Αίγυπτο που πρόσφατα ανακάλυψε μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου. Θα τα στρίξουμε όλα αυτά. Και στο πλαίσιο αυτό, ως μια πρωτοβουλία που ήθελα αμέσως μετά το άτυπο, την άτυπη υπουργική συνάντηση στην Μάλτα, θα έρθουν υπουργοί από τη Βόρεια Αφρική, τη Μεσόγειο και το Ισραήλ Καθώ και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα συναντηθούν λοιπόν όλοι αυτοί για να συζητήσουμε τις διάφορες μεθόδους, τι τρεις μεθο... μεσογειακές πλατφόρμες που είναι υποσυζήτηση, ανανεώσιμες και ενεργειακή απόδοση, ε, φυσικό αέριο και φυσικά παραγωγή ενέργεια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα στοιχεία μας. Από πού συλλέγουμε τις στατιστικές μας, ε, αλλά καταλαβαίνω αυτό που μας είπατε για τις τιμές στη Σκανδιναβία και σε ένα βαθμό αυτό που θέλαμε να κάνουμε θα είναι να υπάρχει περισσότερη συνδεσιμότητα ούτω ώστε οι θετικές τιμές, οι χαμηλές τιμές σε ορισμένα τμήματα της Ευρώπης να περάσουν και σε άλλες περιοχές. Παράλληλα βέβαια θα υπάρξουν και κάποιες ενεργειακές απώλειες. Το δικό μου κράτος για παράδειγμα έχουμε μια σύνδεση με την Σικελία από το 2015 και η σύνδεση αυτή λειτουργεί, ορισμένε φορές έχουμε κάποιε διακοπές, αλλά η σύνδεση μεταξύ της Ιταλίας και της Σικελία δεν είναι τόσο καλής διάσταση. υπάρχει πολλή συμφόρηση. Αν βελτιωθεί αυτή η σύνδεση θα αποφελούμεθα και εμεί και θα είχαμε καλύτερες τιμές. Αλλά καταλαβαίνω τι εννοείται κύριε Τουρμα. Η κυρία Ντάλη ε, είπε ορισμένα πολύ σωστά αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στην Μάλτα. Περνάμε λοιπόν από πολύ πιο βαριά παράγωγα του πετρελαίου στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια έγινε αυτή η αλλαγή. Αυτό είχε ως επίπτωση και μείωση των τιμών και 50% μείωση των ε, ρηπαντών και κλείσαμε ορισμένες ε, ιδιαίτερα ρηπογόνες εγκαταστάσεις παραγωγής. Άρα έχουμε συγκεκριμένη επίπτωση στη ζωή των πολιτών. Και θα συνεχίσουμε και άλλες πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο. Θα αντικαταστήσουμε τη μονάδα υγροποιημένου με έναν αγωγό. Τώρα για την ευρωπαϊκή διάσταση. Η ασφάλεια προμήθειας σε φυσικό αέριο. Έχει τρεις πλευρές ε, αυτή η προσπάθεια, συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλεγγύη. Νομίζω ότι τα απορίσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου είναι θαρρυντικά. Υπάρχουν κάποια θέματα που προσπαθούμε να καλύψουμε κάποιες αδυναμίες Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από ομάδε εργασία που συνεδρίασαν τις τελευταίες εβδομάδες, στόχος μας είναι, κατά τη διάρκεια της προεδρίας όχι μόνο να ξεκινήσει η συζήτηση με το Κοινοβούλιο, αλλά και να καταλήξει νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αλλά και συμβολική αυτή η προσπάθεια, αυτό το νομοθέτημα που επηρεάζει την καθημερινότητα. Ο κύριος Ηλικιώτης επίσης έθεσε κάποια θέματα για την ενεργειακή φτώχεια και η κυρία Γκρίφιν έθιξε κάποια θέματα παρόμοια. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα θέμα που μας αφορά. Θα αντιμετωπιστεί μέσω του πακέτου για την καθαρή ενέργεια Θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά στο πακέτο αυτό υπάρχει ο ορισμός των ευπαθών καταναλωτών. Πρώτο βήμα. Ίσως δεν επαρκεί, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Πρέπει να το προωθήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Και φυσικά είναι τμήμα της συζήτησης του πακέτου. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Γιατί και η κυρία Γκρίφιν και η κυρία Ντάλι τόνισαν ότι, τα θε... ότι οι πολίτες δεν πρέπει να επιλέγουν ανάμεσα στη θέρμανση και την ε, διατροφή τους. Συμφωνούμε απόλυτα. Και η κυρία Γκρίφιν βεβαίως ε, έχει αναλάβει συγκεκριμένες δραστηριότητες και της εύχομαι κάθε επιτυχία από την ε, εκδήλωση αυτή στην Γάνδη. Ο κύριος Ηλικιώτης επίσης έθεσε ερωτήματα για τη Μάλτα ότι είμαστε απομονωμένοι από το δίκτυο. Είναι γεγονός. Τώρα έχουμε αυτή την σύνδεση με την Σικελία που μας δίνει περίπου 200 μεγαβατόρες, μια μικρή χώρα, πρέπει να έχει ενεργειακή ασφάλεια. Αν λοιπόν ο μεγαλύτερος κινητήρας αυτού, αυτής της σύνδεσης ε, αντιμετωπίσει προβλήματα, έχουμε επαρκή αποθέματα ενέργειας για να συνεχιστεί η παροχή ρεύματος στη χώρα. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα ενέργεια που βασίζεται πρώτα απ' όλα στις ανανεώσιμες, στη Μάλτα το καθαρό αέριο, και επιπλέον και μία λύση σε περίπτωση που θα έχουμε προβλήματα με το βασικό μας μείγμα και θέλουμε οπωσδήποτε η Κομισιόν να προωθήσει περαιτέρω τέτοιες πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν ότι κάθε κράτος μέλος είναι σωστά διασυνδεδεμένο. Επίσης ο κύριος Ηλικιώτης αναφέρθηκε στην ε, διάσταση της Ανατολικής Μεσογείου και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ με αυτές τις ε, ε, πρόσφατες ε, ανακαλύψεις θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο κοντά στην Κύπρο είναι πιο εύκολο να προωθήσουμε την περιφερειακή συνεργασία εδώ και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Το 2014 μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Κυπριακή Κυβέρνηση οργανώσαμε μια κοινή εκδήλωση στη Μάλτα για να ξεκινήσει η διαδικασία η Ευρωμεσογειακή και οι Ιταλοί διοργάνωσαν κάποια περαιτέρω εκδήλωση για το θέμα αυτό στη Ρώμη. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια μέσω τη εκδήλωση στην Μάλτα τον Μάιο. Θα πιέσουμε για να υπάρξει μια ευρωμεσογειακή πλατφόρμα όχι μόνο για το αέριο αλλά και για τις ανανεώσιμες και γενικά για την παραγωγή ενέργειας. Να απαντήσω τώρα στην κυρία Κάπελ που αναφέρθηκε στις προτάσεις που υπέβαλε ο κύριος Σεύκοβιτς και ο κύριος Κανιέτε για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους Προφανώς θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να υπάρξει η αναγκαία δυναμική για να προωθηθούν τα θέματα αυτά κατά την Προεδρία μας. Προφανώς τα 28 κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή μελετούν αυτές τις προτάσεις. Είναι τεράστιο διαστάσεων νομοθεσία, διακυβέρνηση, ανανεώσιμες, αποδοτικότητα, σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρισμού και διάφορα άλλα στοιχεία. Κρίσιμα αυτά για να υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στην Ευρώπη και φυσικά θα προωθήσουμε αυτό το θεματολόγιο. Τα κράτη-μέλη μα ζήτησαν όμω κάποιο χρόνο για να μελετήσουν ε, όλα αυτά τα έγγραφα και έχουμε δεσμευθεί ότι θα τα ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα του πακέτου κατά την Προεδρία μας. Θέλουμε να υπάρξει πραγματικά έντονος ρυθμός και έχουμε προσθέσει και συνεργάτες στη μόνιμη αντιπροσωπεία για να καταστεί δυνατό. Έχουμε συνεδρίαση μίας ομάδας εργασίας κάθε εβδομάδα για ενεργειακά θέματα άρα περίπου τέσσερι συνεδριάσεις τέτοιε το μήνα και θα αυξήσουμε τον αριθμό. Θέλουμε να υπάρχουν δύο τέτοιε συνεδριάσει ε, περαιτέρω για να έχουμε έξι το μήνα. Μόνο έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να διατηρηθεί αυτό ο ρυθμός και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ, θεωρούμε ότι η γενική προσέγγιση για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, αυτά τα δύο νομοθετήματα που είναι τα πιο εύκολα να προωθηθούν για να επιτύχουμε ε, ταχεία συνένεση. Τώρα θα ανοίξουμε και τα άλλα. Τώρα η οδηγία για την ε, αγορά ηλεκτρισμού είναι πολύ δύσκολη ορισμένη, ανησυχούν για τον άνθρακα και για τον μηχανισμό διασφάλισης. Θέλουμε λοιπόν το πακέτο αυτό να είναι ο κατάλληλος συνδυασμό μέτρων για να προχωρήσουμε, να διατηρήσουμε τον ρυθμό και θα έχω συγκαλέσει ε, συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας το Φεβρουάριο για να δούμε τις απόψει και άλλων κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Κύριε Βέρντερ, είπατε ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στις ανάγκες του κόσμου. Και είπατε πόσο σημαντική είναι η επισήμανση των ενεργειακών προϊόντων. Και σίγουρα πλουστευμένες ετικέτες θα βοηθήσουν ε, το, τους πολίτες να κάνουν τεκμηριωμένες περιστατωμένες επιλογές και να γνωρίζουν και το κόστος των συγκεκριμένων προϊόντων, τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα τεχνικό θέμα που αφορά την εφαρμογή, αν θα εφαρμόσουμε καταξιοδότηση, εφαρμοστική πράξη και εκεί υπάρχουν κάποιες τριβές και εντάσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το ποιο είναι το καταλληλότερο μέσο, αλλά ε, θα έχουμε και άλλα θέματα που θα επηρεάσουν τη συγκεκριμένη συζήτηση. Εγώ πάντως θα καταβάλω προσπάθειες να τα διεκπαιρεώσουμε κατά τη διάρκεια της δική μας Προεδρίας, βρίσκοντας τη σωστή συνένεση, γιατί είναι θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συμπολιτών μα. Ο κύριος Κόχλιτσεκ με ρώτησε ποιο είναι το μείγμα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στη Μάλτα. Ίσως ε, δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας, συγγνώμη. Στην Μάλτα έχουμε κάποιες, ε, κάποιους γεωφυσικούς περιορισμούς και η κυβέρνηση ε, είχε κάποιους ενδιάμεσους στόχους τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχουμε αλλάξει το ενεργειακό μας μείγμα. Αρχικά η προηγούμενη κυβέρνηση επικεντρωνόταν στην ε, ανεμογεννήτρη, στην αιωλική ενέργεια, αλλά λόγω περιβαλλοντικών λόγων και μεταναστευτικών ροών αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε την αιωλική ενέργεια και να έχουμε στο μείγμα μας αιωλική ενέργεια ε, και χρησιμοποιούμε κάθε ε, οροφή, κάθε ελεύθερο χώρο για να μπορούμε να εγκαταστήσουμε ήλιος στους και να δημιουργήσουμε ε, περισσότερη, να παράγουμε περισσότερη ηλιακή ενέργεια. Επίσης βιοκαύσιμα και έτσι πιστεύουμε ότι θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κυρία Γκρίφη, νομίζω πίνησα στα δικά σας ερωτήματα για τους ευάλωτους καταναλωτές και την ενεργειακή φτώχεια. Με ενδιαφέρει και προσωπικά αυτό το θέμα και θα φροντίσω να περιληφθεί στο πακέτο για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους. Και το θέμα δεν είναι τόσο οι ορισμοί όσο τα μέτρα. Επίσης, τέθηκαν και ερωτήσεις για την προσωπική μου οικονομική κατάσταση από συναδέλφους της αντιπολίτευσης στη Μάλτα. Καταρχήν ε, με συμβούλευσαν να απαντήσω ότι θα πρέπει εδώ να εκπροσωπήσω τα κράτη-μέλη και να αποφύγω συζητήσεις για τα εθνικά ζητήματα. Αλλά από σεβασμό προς τους ευρωβουλευτές θα ήθελα να δώσω κάποιες πληροφορίες και για τα θέματα αυτά. Τα οικονομικά μου θέματα και η οικονομική μου κατάσταση ήταν σαφής. Ε, δημιούργησα ένα οικογενειακό τραστ για να διαχειριστώ κάποια οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία και οικογενειακές μας επενδύσεις. Η εταιρεία αυτή μάλιστα δεν συστήθηκε μετά, το, μετά τις εκλογές του 2013, λάθος. Επίσης, ε, οικειοθελώς ζήτησα φορολογικό έλεγχο για όλα τα οικονομικά μου θέματα, κάτι που είναι άνευ προηγουμένου και κανένα πολιτικό στη Μάλτα δεν είχε ζητήσει κάτι τέτοιο και συνεχίζεται αυτό ο φορολογικό έλεγχο ε, στα οικονομικά μου και μάλιστα ε, καλύπτει όλη μου την οικονομική κατάσταση, όχι μόνο τη συγκεκριμένη εταιρεία και πιστεύω ότι θα ε, αναδεθεί γρήγορα η αλήθεια. Επίση θα γίνει ο έλεγχο και των και τις οικονομικές εταιρείες που συνοδεύει αυτό το οικογενειακό τραστ. Οπότε σας διαβεβαιώ ότι λαμβάνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι και δεν θέλω να περιοριστούμε εδώ στα ενδοκομματικά, ενδοπολιτικά θέματα της Μάλτας. Ήρθα εδώ για να εκπροσωπήσω το Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσουμε σοφά τη Μαλτέζικη Προεδρία με την ενεργειακή επισήμαση που ενδιαφέρει τον κόσμο, με την καθαρή ενέργεια, το SOS για το φυσικό αέριο. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ε, και θα έχουμε ένα καταπληκτικό παραστατικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπλοκο, απαιτητικό, θα απαιτήσει μεγάλη συμβολή των ενδιαφερομένων και κοινοβουλευτικό έλεγχο και προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να διαμορφώσουμε τελικά μια δεσμή μέτρων για ε, ενέργεια σε προσιτές τιμές, καλές διασυνδέσεις, καθαρό αέρα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προώθηση πρώτα απ' όλα της ενεργειακής απόδοσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς, γιατί είναι πραγματικά ιστορική στιγμή, μια και για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε Μαλτέζικη Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία της Προεδρίας σας θα είναι και επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτυχία και της δικής μας Επιτροπής που συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επόμενη μας ε, συνεδρίαση συνεχίζεται αύριο στις 9 το πρωί. Σε τρία λεπτά όμως θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Σε τρία λεπτά συνεδρίαση των συντονιστών στην ίδια αίθουσα και αύριο το πρωί στις 9 συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε.